θεσή του όσον αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, κύριε Σιγητά. Κάποιο τεχνικό πρόβλημα υπάρχει και δεν ακούγεται.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 Non, ça va pas. Ça va pas? Τώρα είναι εντάξει, τώρα είναι εντάξει. Εντάξει είναι τώρα, είναι εντάξει. Τώρα ακούγεται καλά. Τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε. Λύθηκε το τεχνικό πρόβλημα λοιπόν. Συνεπώς έλεγα ότι πήραμε 294 προτάσεις τροποποίησεων. Πρόκειται για πολλές τροπολογίες όπως καταλαβαίνετε, πάρα πολλές. Την τελευταία φορά είπα ότι πρόκειται όντως για 294 τροπολογίες, όμως όσον αφορά την ουσία των τροπολογιών αυτών, υπάρχει μεγάλη σύγκληση μεταξύ πολλών. Και έτσι, όπως το είπα και την προηγούμενη φορά, το ξαναλέω και τώρα, είμαι αισιόδοξο για το τελικό αποτέλεσμα. Είμαι αισιόδοξο γιατί η διαδικασία διαπραγματεύσεων προχώρησε πολύ καλά. Στην αρχή παρουσίασα 24 συμβιβαστικές προτάσεις και μετά πρόσθεσα και άλλες 10. Προσπάθησα να λάβω υπόψη μου και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και όλες τις προτάσεις που πριν από δύο εβδομάδες μου υπέβαλαν οι συνάδελφοι. Σήμερα το πρωί καταφέραμε να ετοιμάσουμε 21 συμβιβαστικές τροπολογίες. Από αυτές τις 21 συμβιβαστικές τροπολογίες καταφέραμε και ελπίζω ότι όντω θα πετύχουμε να έχουμε διακανονίσει όλα τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα, το πρόβλημα ήταν ότι ο καθένας ήθελε να χρησιμοποιήσει τη δικιά του διατύπωση. Άρα χρειάστηκε μεταξύ μας να καθίσουμε και να ερμηνεύσουμε λιγάκι τις λέξεις για να καταλήξουμε σε ένα νόημα. Γλωσσικό δηλαδή ήταν το ζήτημα σε πάρα πολλές περιπτώσεις αλλά υπήρξαν και άλλα προβλήματα που έπρεπε να λυθούν. Προβλήματα που είχαν να κάνουν κυρίως με το περιεχόμενο των κατευθυντηρίων γραμμών. Δηλαδή, τι έπρεπε να συμπεριληφθεί στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές. Εννοείται ότι συζητήσαμε επί της ουσίας, αλλά τελικά καταφέραμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Σε ποιο πεδίο Πολλοί είπαν για τα επόμενα δέκα χρόνια πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι, να έχουμε φιλόδοξους στόχους. Αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε και πέρα από τα δέκα χρόνια. Οπότε ο κύριος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η πλήρης απασχόληση. Σε δέκα χρόνια ή μετά τα δέκα χρόνια. Για μένα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για να βρω μια διατύπωση που να κάνει του στόχου που είναι η πλήρης απασχόληση σε 10 χρόνια, το 2, σε 10 χρόνια από τώρα. Ακόμα κι αν προς το παρόν οι κατευθυντήριες γραμμές είναι για τρία χρόνια. Όμως θέλαμε να εκφράσουμε το στόχο μας σε 10 χρόνια ή και αργότερα. Τώρα υπήρξε κάποια απόκληση απόψεων βέβαια για ορισμένα ζητήματα όσον αφορά την απασχόληση. Μιλάμε για την πλήρη απασχόληση, μιλάμε για την ποιότητα της απασχόλησης. Αν έπρεπε να μιλήσουμε για την ποιότητα, αν έπρεπε να μιλήσουμε για τις καλές θέσεις απασχόλησης ή όχι. Τελικά, τελικά καταλήξαμε να υιοθετήσουμε την πρόταση του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας για την αξιοπρεπή εργασία, decent work. Έτσι λοιπόν συμπεριλάβαμε την έκφραση αυτή αξιοπρεπής εργασία στην ε, πρότασή μας. Επίσης, εμείναμε και στην ιδέα της ίδιας εργασίας για ίδιο μισθό. Και θελήσαμε να δούμε κατά πόσο ο ελάχιστος μισθός ως έννοια είναι κάτι που υπάρχει σε όλες τις χώρες. Γιατί γνωρίζουμε ότι σε ορισμένες χώρες ο ελάχιστος μισθός δεν υπάρχει σαν έννοια ακόμα. Και μια που μιλάμε για κοινέ πολιτικές όπου τα κράτη-μέλη όμως έχουν την ευχέρεια να θέσουν σε εφαρμογή τις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, το ζήτημα αυτό διακανονίστηκε. Έρχομαι τώρα στο ευρώ. Ποιος είναι ο ρόλος του ευρώ στην τελική μορφή του συμβιβασμού μας. Ε, λοιπόν, δεν μιλάμε πια για το ρόλο του ευρώ εκεί. Έπρεπε να κρατήσουμε την προστασία των θέσεων απασχόλησης, που ήδη υπάρχουν. Δεν θέλουμε να μιλάμε δηλαδή μόνο για τις θέσεις εργασίας που θέλουμε να δημιουργηθούν, αλλά και για τη διατήρηση εκείνων που ήδη έχουμε. Και όλα αυτά χρειαζόταν συμβιβασμοί. Δεν πρέπει επίσης να μειωθεί ο διαρθρωτικός, ε, ε, η ανεργία μόνο, αλλά να πάμε ακόμα παραπέρα. Και αυτή η ιδέα παραμένει στο συμβιβασμό. Τελικά μπόρεσα να δεχτώ όλες αυτές τις προτάσεις. Για μένα Πρόκειται για μια αισιόδοξη πρόταση. Οι σοσιαλιστές συνάδελφοι έκαναν την εξής πρόταση. Θέλανε να δούνε όχι μόνο στόχους, αλλά και υποκατηγορίες στόχων στο κείμενο. Οπότε φτιάξαμε και τέτοιες κατηγορίες στόχων που είναι οι εξής. Απασχόληση νέων, ατόμων 60 με 65 ετών, απασχόληση για τα άτομα με αναπηρίες, για μετανάστες νόμιμους. Όλες αυτές οι κατηγορίες στόχων έχουν ως αντικείμενο την μείωση κατά 10% της ανεργίας. Για μένα αυτές οι υποκατηγορίες είναι πολύ φιλόδοξες. Όμως ο τελικός μας στόχος ποιος είναι. Είναι να δώσουμε μια όθηση στα κράτη-μέλη προκειμένου να κάνουν πραγματικές προσπάθειες για να μειωθεί η ανεργία. Οπότε, τελικά, εφόσον αυτό είναι ο κύριος στόχος μας, γιατί να μην βάλουμε και τέτοιες υποκατηγορίες στόχων μέσα στις συμβαστικές τροπολογίες. Έρχομαι τώρα στην ανάγκη που υπάρχει για κατάρτιση και επιμόρφωση. Εδώ οι συνάδελφοι τόνισαν όλος ιδιαιτέρως το ότι δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τις ανάγκες της βιομηχανίας, αλλά πρέπει να κοιτάμε και τις ανάγκες της οικονομίας. Και έτσι να αποφασίζουμε για την κατάρταση και την επιμόρφωση. Τέλος, οι ίσες ευκαιρίες και η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών περιλαμβάνεται στις συμβαστικές μας τροπολογίες. Από εκεί και πέρα θα δούμε οι συνάδελφοι πώς θα αντιμετωπίσουν τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Πάντως εγώ πιστεύω ότι μέσα από τις 21 αυτές συμβιβαστικές τροπολογίες ειλικρινά όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να βρουν τις επιθυμίες τους και έτσι μπορούν να τις υποστηρίξουν. Ελπίζω ότι θα υπερψηφιστούν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν με ένα τιτάνιο έργο. Πραγματικά η δουλειά ήταν πάρα πολύ μεγάλη προκειμένου να ετοιμαστούν οι συμβαστικές αυτές τροπολογίες. Ευχαριστώ επίσης και όλους τους κοιόδης εισηγητές από όλες τις πολιτικές ομάδες. Χάρη στην συνεργασία όλων των σκιωδών εισηγητών, καταφέραμε να φτάσουμε σε αυτό το καλό αποτέλεσμα. Ελπίζω ότι το αποτέλεσμα θα ικανοποιήσει όλους και θα το στήριξετε. Για άλλη μια φορά, ευχαριστώ πολύ και παρακαλώ όλοι αύριο να στηρίξετε τις συμβαστικές αυτές τροπολογίες στη στιγμή της ψηφοφορίας. Έτσι θα έχουμε κάνει ένα βήμα προς τα μπρος και θα έχουμε μια σημαντική και ισχυρή θέση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέναντι στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Περιμένω τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε. Η κυρία Στένρουτ και μετά κυρία Τσουβινού. Ευχαριστώ ε, κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο έρη ως εισηγητή, ο οποίος ε, πραγματικά κατόρθωσε ε, αντίθετες θέσεις να τις συμπεριλάβει σε ένα συμβασμό. Ευχαριστώ και τους άλλους συζητητές. Εγώ θεωρώ ότι η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Αγωνιστήκαμε σκληρά για να συνάψουμε τους συμβασμούς και θέλω να ελπίζω αύριο στην Επιτροπή να διαμορφωθεί η σωστή πλειοψηφία. Για μα, για τη δική μα την πολιτική ομάδα, ήταν πολύ σημαντικό να υπάρξει σαφής ορισμός αυτού που εμεί κατανοούμε ως καλή εργασία ε, στις κατευθυντήριε γραμμές ε, περί απασχόλησης. Ε, να απαγορεύεται το dumping στους μισθού, ο στόχο για την πλήρη απασχόληση να μην χαθεί. Αυτά για μα ήταν εξίσου σημαντικά όπως και το να επιτύχουμε τους ενδιάμεσους στόχους μας ε, μέχρι το 2014 γιατί θεωρούμε ότι το 2020 είναι πολύ μακριά, ως εκ τούτου θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να ε, εξετάσουμε ενδιάμεσα κατά πόσο ο δρόμος είναι σωστός, μήπως χρειάζονται βελτιώσεις, πολύ σημαντικά όλα αυτά. Όπως επίσης και η συμπερίληψη των κοινωνικών εταίρων ε, και όλων των εμπλεκομένων στην ε, εκπόνηση νομολογίας. Θα μπορούσα να αναφέρω πάρα πολλά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα περιοριστώ στο να πω καταρχήν ευχαριστώ πολύ για την πολύ καλή συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Όρη. Όπως θα διαπιστώσετε όλοι κάναμε πολλούς συμβιβασμούς εδώ δεν θεωρώ ότι είναι τέλειο, αλλά είναι ένα συμβιβασμό. Για κανέναν από εμά δεν είναι τέλειο το αποτέλεσμα, αλλά αυτή είναι η πολιτική άλλωστε. Ε, φαντάζομαι ότι θα μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε το κείμενο αύριο. Και αυτό που έχει σημασία για μα ω Επιτροπή είναι ότι υπάρχει κάποιο επιπρόσθετο όφελο ε, σε αυτά που μα λέει το Συμβούλιο και επίση ενισχύει το κείμενο το οποίο μας έχει δοθεί. Το ενισχύει σε θέματα διακυβέρνησης, σε θέματα αξιοπρεπούς εργασίας, σε θέματα φύλου. Είναι πιο ισορροπημένο, ε, έχει μια πιο ισορροπημένη εικόνα για το flexicurity και από πλευράς μας, δεν, ναι, δεν συμπεριλαμβάνεται στο συμβιβασμό, αλλά ε, ελπίζουμε να μπορέσετε να υποστηρίξετε και τις ε, δικές μας προτάσεις αύριο και να τις συμπεριλάβουμε και αυτά στις κατευθυντήριες γραμμές. Θεωρούμε ότι έχουμε πολλά να προσθέσουμε στο κείμενο του Συμβουλίου και αυτό το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό είναι αυτό το σχετικό στόχος του 10% για τις ειδικέ ομάδες διότι πρόκειται για τις πλέον ευάλωτες ομάδες, ε, νέοι άνθρωποι, μετανάστες και ούτω καθεξής και στοχεύοντας αυτούς ε, με αυτό το 10% ε, θεωρώ ότι μπορούμε να επιτύχουμε κάτι. Υπάρχει η διάσταση της δημιουργίας θέσεων εργασίας και συμπερίληψη στην αγορά εργασίας. Ε, να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους συναδέλφους και ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε τουλάχιστον να περάσουμε την άποψή μας προς το Συμβούλιο. Ο κύριος Μαν. και μετά η κυρία Κορνέλσεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι ο κύριος Ερή ε, πέτυχε την συνένεση εκείνων που εργάστηκαν για την έκθεση και κυρίως εργάστηκαν για τους συμβιβασμού. Είναι λοιπόν ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο. Η κυρία Τουμούν είπε ότι δεν είναι τέλεια η έκθεση, ε, καλή είναι. Σημασία έχει ότι καταλήξαμε σε συμβιβασμό ε, κάναμε παραχωρήσεις και οι δύο πλευρές. Βεβαίως ε, υπάρχουν ακόμα ίσως κάποια ερωτηματικά. Αυτά σε σχέση με τον ILO. Ε, ποια είναι η καλή δουλειά η ποσότητα και η ποιότητα, αυτά είναι καθοριστικής σημασίας. Εκείνο που παίζει ρόλο είναι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι αυτός τουλάχιστον είναι ένας συμβασμός που είναι πολύ σημαντικός γιατί έχει άμεση σχέση με την πραγματικότητα. Πολλές εκθέσεις ε, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας ε, ε, αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που δημιουργήσαμε μια κοινώ αποδεκτή βάση. Το θέμα της, του δίκαιου μισθού, του dumping, θεωρώ ότι μπορούμε βέβαια να τσακωθούμε για τον ορισμό όλων αυτών των όρων στις γλώσσες μας εγώ όμως πιστεύω ότι τελικά ε, η κατεύθυνση είναι σωστή. Βεβαίως και υπάρχουν αποχρώσεις κατά την εφαρμογή στις διάφορες χώρες. Σημασία έχει να λέμε ότι όποιος εργάζεται πρέπει να αμείβεται και να μπορεί να ζει, όχι να επιβιώνει. Αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο. Και ήθελα επίσης να επισημάνω ότι υπάρχει ένα θέμα ε, το οποίο είναι κάπως κρίσιμο και δεν αφορά την έκθεση ΕΡΗ. Πρόκειται για το ε, τι θα γίνει τελικά με τις ε, ποσοστώσεις. Εχθές και σήμερα ε, είχαμε την ευκαιρία να συναντηθούμε με μέλη του Γερμανικού Κοινοβουλίου, του Bundestag και η Πρόεδρός μας ήταν παρούσα. Και αυτοί λοιπόν θεωρούν ότι ε, βεβαίως και παίζει ρόλο το μακρόπνο πρόγραμμα, αλλά πρέπει και ενδιάμεσα να κάνουμε κάποιες επανεξετάσεις. Το θέμα των ποσοστώσεων αντιμετωπίζεται λίγο διαφορετικά στα κράτη-μέλη, ε, γιατί Μερικοί λένε, αν δηλαδή έχει ικανοποιηθεί η ποσόστοση, τι θα γίνει μετά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αρχίσει να βαθμολογεί τις διάφορες χώρες. Κάποιες, ε, κάποιοι λένε ότι εμείς δεν θα δεχθούμε την αξιολόγηση. Για μένα λοιπόν αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη για να μπορούμε να μετακινηθούμε προς τα εμπρός, να πούμε ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τον προσανατολισμό στην ε, ποιότητα και πρέπει να μειώσουμε τον αριθμό των νέων που εγκαταλείπουν το σχολείο γιατί οι άνθρωποι δεν θα μπορέσουν να βρουν δουλειά αν δεν πληρούν κάποια κριτήρια και τα κριτήρια αυτά γίνονται και πληρούνται μέσα από την εκπαίδευση. Εκεί λοιπόν πρέπει να επενδύσουμε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ωρί και όλους τους άλλους που εργάστηκαν για την έκθεσή του ως ασκιώδης εισηγητές. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορνέλισον και μετά ο κύριος Έλμερ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω και τον κύριο και όλους τους κοιόδης εισηγητές για την ε, τεράστια δουλειά που έκαναν. Πράγματι, οι τροπολογίες ήταν πάρα πολλές και περάσαμε πάρα πολύ χρόνο συζητώντας για αυτές και διαπραγματευόμενοι. Νομίζω ότι η δουλειά όμως μόλις ξεκινάει με την αυριανή ψηφοφορία. Ελπίζω ότι θα έχουμε μεγάλη πλειοψηφία και στην Ολομέλεια. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε το Συμβούλιο να καταλάβει. Αν δούμε την αρχική πρόταση και την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, διαπιστώνουμε ότι το Συμβούλιο έχει αλλάξει τρεις λέξεις. Δηλαδή, μόνο τρεις λέξεις άλλαξε μετά από όλες τις αλλαγές που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι σημαίνει αυτό ότι όλη αυτή τη δουλειά την κάναμε για τρεις λέξεις. Ε, όχι. Αυτή τη φορά ελπίζω το Συμβούλιο να μας, πάρει, να μας λάβει υπόψη και εμάς και τις παρατηρήσεις μας. Ο κύριος Έλμερ και μετά Μωρά. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω με τη σύρια μου τον κύριο Όρη, διότι ανέλαβε ένα Ηράκλειο έργο, όπως το ανέφερε και ο ίδιος. Πόσοι από τους συναδέλφους μας σήμερα έχουν συζητήσει τα θέματα αυτά με τους εργοδότες και όχι μόνο με όσους εργάζονται στα θεσμικά όργανα. Εγώ έχω μιλήσει πολύ με εργοδότες και διαμαρτύρονται για το την υπερβολική νομοθεσία σε θέματα απασχόληση που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεχώ νέε ρυθμίσει που είναι πάρα πολύ δαπανηρέ και είναι πολύ δύσκολο να επιβιώσει κάποιο με αυτέ τι ρυθμίσει. Ποιο είναι αυτό ο οποίο αποφάσισε ότι πρέπει να έχουμε κατευθυντήριε γραμμέ. Ε, άκουσα τον κύριο Όρη να λέει ότι είμαστε 10 χρόνια μπροστά. Αυτό νομίζω ότι θριαμβεύει η ελπίδα και όχι η πείρα. Θα θυμάστε την ε, στρατηγική τη Λισαβόνα, η οποία ναι, μεν υποτίθεται ότι έβλεπε 10 χρόνια μπροστά και τελικά πέτυχε παταγωδό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε το 2020 και τη διαδικασία αυτή και πάρα πολλοί προβλέπουν ότι δεν θα πάει και πολύ καλύτερα με τη, από τη στρατηγική τη Λισαβόνα. Να θέσουμε στόχου. Όσου στόχου και να θέχουμε, ε, αν δεν προσπαθήσουμε να του επιτύχουμε, θα παραμείνουν κενό γράμμα. Έχουμε το στόχο τη πλήρου απασχόληση και αυτό είναι πάντα το ιδεώδε, είναι πάντα το όνειρο. Ε, εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε, αν υπήρχε πλήρη απασχόληση, Όμω θα είχαμε μια πολύ στατική και καθόλου ευέλικτη αγορά εργασία και αυτό φυσικά δεν θα ήταν καλό για την οικονομία. Σαφώ είναι επιθυμητό αυτό ο στόχο, αλλά δεν ξέρω πόσο αποφασισμένοι είμαστε να τον επιτύχουμε. Μιλάμε για τις διαφορές μεταξύ της δημιουργίας θέσεως εργασία και της διασφάλισης των θέσεων εργασία. Από τη δική μου την πείρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά από τα κράτη-μέλη εστιάζουν σχεδόν αποκλειστικά στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας και όχι στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Θέλουν ε, δηλαδή να κάνουν την αγορά λιγότερο ευέλικτη, οι ε, εργοδότε δεν είναι διατεθειμένοι να ε, προσλάβουν περισσότερους εργαζόμενου και φυσικά οι προοπτικές για την απασχόληση είναι μάλλον δύσκολε. Υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας. Οι πράσινες θέσεις εργασίας είναι εφήμερες και συνήθως κάθε πράσινη θέση εργασίας που δημιουργείται καταστρέφει δύο θέσεις εργασίας σε άλλους τομείς, καταστρέφοντας πολύ αποτελεσματικές θέσεις. Κάποιοι αναφέρθηκαν στην αφαίρεση του ευρώ από την έκθεση. Ε, εμένα με χαροποιεί το γεγονό αυτό, διότι κάποιοι λένε ότι το ευρώ είναι αυτό το οποίο προσθέτει σταθερότητα στην ευρωζώνη. Από αυτά που βλέπουμε του τελευταίους ε, μήνε, βέβαια, νομίζω ότι είναι απλώ μεταθανάτια ερανή αυτό. Το ευρώ ε, που θεωρείται η κορονίδα της μακροοικονομικής σταθερότητας μάλλον κοιμάται τα τελευταία δύο-τρία χρόνια. Αυτό που επιτυγχάνουμε κυρία Πρόεδρε, εάν επιτυγχάνουμε κάτι ουσιαστικά, είναι να διαφυλάσσουμε τις θέσεις εργασίας των Ευρωβουλευτών που ακούσαμε ότι ε, χρειάστηκαν πάρα πολύ χρόνο να ετοιμάσουν αυτή την ε, έκθεση. Να σας πω την άποψή μας. Νομίζω ότι κανείς εκτός αυτής της αίθουσας δεν θα δώσει σημασία στη δουλειά του κυρίου Όρη. Ε, πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω μιλώντας ειλικρινά, λέγοντας τις σκέψεις μου για την έκθεση αυτή, της οποίας ηγήθηκε ο κύριος Σωρή, αλλά για τη δουλειά που κάνανε και οι σκιώδεις εισηγητές, γιατί από ό,τι κατάλαβα είναι μια συλλογική δουλειά αυτή. Που βοηθάει να βελτιωθεί κατά πολύ το αρχικό κείμενο. Αυτό που μου αρέσει λοιπόν σε αυτή τη δουλειά και που θέλω να υπογραμμίσω όλος ιδιαίτερος είναι από τη μια μεριά έχουμε καταλήξει σε ένα όραμα για το 2020 τι θα γίνει με την απασχόληση δηλαδή τότε σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά συγχρόνως και παράλληλα και έτσι απαντάω στον κύριο Έλμερ νομίζω ας μου επιτρέψει έχουμε διάμεσους στόχους ο Τόμας Μαν πριν αναφέρθηκε σε ποσοστώσεις, σε ποσοτική έκφραση. Αν λοιπόν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους μας για τις κατευθυντήριες γραμμές στην απασχόληση, χρειάζεται μια καθοδήγηση με διάμεσους στόχους, αλλά και ανά σημείο. Όχι γενικά μόνο στην Ευρώπη και πιο τοπικά. Νομίζω λοιπόν ότι οι υπεύθυνοι σε περιφερειακό επίπεδο, πολιτικά και οικονομικά, συμφωνούν με τη στρατηγική μας αυτή. Δεύτερον, φυσικά και μπορούμε να γράψουμε ό,τι κατευθυντήριες γραμμές θέλουμε για την απασχόληση. Αν όμως δεν ξεκινήσουμε με το σύστημα εκπαίδευσης, προκειμένου να βγαίνουν ε, νέοι με προσόντα που να είναι χρήσιμα, δεν θα έχουμε κάνει τίποτα. Γιατί το να βγαίνουν νέοι χωρίς τα κατάλληλα προσόντα μπαίνουν στο περιθώριο και μετά είναι χαμένοι. Διότι για να μπει κανεί στην αγορά εργασία, εννοείται ότι πρέπει να έχει κάποια προσόντα. Α φροντίσουμε λοιπόν να το πετύχουμε αυτό πρώτα απ' όλα. Τρίτον, οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές και η συνένεση την οποία πετύχατε από κοινού δείχνει ότι σήμερα έχουμε μια συγκεκριμένη διακυβέρνηση μαζί με τους κοινωνικούς εταίρους. Δεν έχουμε πια όπως παλιά ε, την στάση εκείνη που ή που ήμασταν επικεντρωμένοι στην επιχείρηση ή που είμαστε επικεντρωμένοι στους εργαζόμενους. Όχι, τώρα λαμβάνουμε υπόψη μας και τα συμφέροντα τη επιχείρηση στον κόσμο οικονομία στον οποίο ζούμε, αλλά και την εξέλιξη των εργαζόμενων με την διαβίω κατάρτιση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο στοιχείων μπορεί να μας βοηθήσει να πετύχουμε με τις κατευθυντήριες γραμμές μας για την απασχόληση. Όντως πρέπει οι άνθρωποι εργαζόμενοι να μπορούν να προσαρμοστούν στις ανάγκες της ζωής, της επιχείρησης. Άρα δεν πρόκειται μόνο για υψηλά προσόντα, πρόκειται για συνδυασμό της δυναμικής των επιχειρήσεων και των δυνατοτήτων των εργαζομένων. Αυτά τα δύο πρέπει να τα συνδυάσουμε και έτσι να προχωρήσουμε με τις κατευθυντήριες γραμμές βάσει των στόχων μας. Ευχαριστώ. Η κυρία Οβίρ και μετά η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σκιώδη συγητή εκ μέρους των φιλελευθέρων. Πράγματι ήταν μια πολύ καλή δουλειά και θα ήθελα να επενέσω κυρίως τον τρόπο με τον οποίο κατόρθωσε να μας πείσει. Γιατί όπως και όλοι οι άλλοι και εγώ πιστεύω ότι υπήρχαν πάρα πολλά που έπρεπε να ληφθούν υπόψη. Έχουμε 27 κρατημέλη, την οικονομική κρίση. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ε, ενδείξεις ε, ότι ε, φεύγουμε από την κρίση και φάνηκε κάποια στοιχεία ανάκαμψης, βέβαια με υψηλή ανεργία. Πρέπει ως εκ τούτου οπωσδήποτε να αυξήσουμε τις ε, θέσεις εργασίας, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να βρουν απασχόληση. Από τις 294 ε, τροπολογίες εμείς ε, πετύχαμε 21 συμβιβαστικές. Ε, αυτό ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε. Ίσως ε, να κατατεθούν και κάποιες άλλες καλύτερες. Με πάση περιπτώσει κάναμε ό,τι μπορούσαμε και πραγματικά ελπίζουμε ότι τελικά δεν θα αποτύχει αυτό το πρόγραμμα. Αν δεν κάνουμε τίποτα. Ούτε εμείς, ούτε τα κρατημέλη, προφανώς θα παραμείνουμε στάσιμοι. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να επιτρέψει τον εαυτό της τέτοια πολυτέλεια. Γι' αυτό λοιπόν εύχομαι καλή τύχη στον εισηγητή κατά την διαδικασία έγκρισης της εισήγησής του. Η κυρία Όρκεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Ρή. Δεύτερον, να πω ότι πραγματικά είναι μια πολύ φιλόδοξη έκθεση και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να συμπεριλάβει πολλέ και αντικρουόμενε απόψει. Όχι αν θέλετε ακριβώ αντικρουόμενε, εν πάση περιπτώσει έχει γίνει πολλή δουλειά πάνω σε αυτέ. Ε, συμφωνώ με κάποιον συνάδελφο που είπε ότι είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Πάντω τα σημαντικότερα θέματα εξετάστηκαν. Ο κύριο Μαν λέει ότι πρέπει πρέπει να δούμε λιγάκι το θέμα των ορισμών ε, και εγώ έχω εδώ ένα κατάλογο ορισμών. Ε, θα τον δώσω στη γραμματεία για να σας τον διανύμει, γιατί όταν μιλάμε για κάποια πράγματα πρέπει όλοι να έχουμε συμφωνήσει το εννοούμε ακριβώς το ίδιο. Ε, τώρα, αυτό που δεν μου αρέσει πολύ στην έκθεση είναι ότι υπάρχουν αρκετές επαναλήψεις, αλλά δεν θα αναφερθώ λεπτομερώς σε αυτά. Ε, να πω όμως κάτι πιο συγκεκριμένο. Στην συμβαστική πρόταση I, ε, λατινικό, εκεί θα πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο για την ε, αντιμετώπιση, την αποτελεσματική των διακρίσεων. Και υπάρχουν ένα-δύο άλλο θέματα στην συμβαστική πρόταση N, Εκεί γίνεται λόγος για τον ανταγωνισμό. Δεν είμαι σίγουρη ότι αυτό είναι συμβατό με, τον, με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Μιλάμε επίσης για το ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να αναθεωρήσουν τα φορολογικά του συστήματα. Το review μπορεί να μείνει, δεν είναι και ιδιαίτερα ισχυρό. Και ένα σχόλιο για τη συμβαστική πρόταση P, όπου λέμε ε, να πληρούνται οι όροι σε ορισμένες ε, θέσεις απασχόλησης. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι θέσεις απασχόλησης, αλλά ίσως μπορεί να μας το εξηγήσει ο κύριος ε, Όρη. Οι περισσότερες απόψεις αναφέρονται και συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Κορνέλισον ότι πράγματι το Συμβούλιο πρέπει να μας λάβει περισσότερο υπόψη τους τώρα από ό,τι κατά το παρελθόν και ελπίζω να το πράξουν αυτό. Πρόεδρε, ε, κοιτάξτε, θέλω να πω ότι οι σκιώδεις ηγητές και οι βοηθοί εργάστηκαν πάρα πολύ σκληρά για την έκθεση αυτή και ορισμένοι συνάδελφοί μου με ενημέρωσαν με την ένταση ε, με την οποία έγιναν συζητήσει, οι οποίε βέβαια αποτύχθηκαν επικοδομητικές. Εμείς ως πολιτική ομάδα θα στηρίξουμε αρκετές από τις συμβαστικές τροπολογίες. Κάποιες, ε, κάποια άλλα εδάφια στο αιτιολογικό ε, θα τα καταψηφίσουμε. Δύο θα αναφέρω που έπαιξαν ρόλο στη συζήτηση. Το πρώτο θέμα αφορά στους στόχους. Υπάρχει μια παλιά αρχή που λέει ότι όποιος δεν γνωρίζει το στόχο πολύ συχνά δεν βρίσκει και το δρόμο. Σε πάρα πολλούς ε, στόχους υποδιατύπωση η έκθεση αυτή ε, παραμένει ασαφής. Εμείς λοιπόν ε, θα επιθυμούσαμε και προτείναμε να συγκεκριμενοποιηθούν κατά τη στόχη. Δεύτερον, η έκθεση αυτή ε, για τα δικά μας τα γούστα ακολουθεί πάρα πολύ αυτή τη σκέψη την γνωστή περί flex security ευελιξίας και ασφάλειας. Ναι, μεν έχει υπήρξει, υπάρξει κάποια πρόοδος, όμως ε, τα συνδικάτα λένε να αλλάξουμε τον όρο και να μιλάμε για securability, δηλαδή να επιμείνουμε περισσότερο έτσι ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια. Ε, κατά την άποψή μας όμως αυτός όρος, αυτή η έννοια δεν εμφανίζεται παρκώ στην έκθεση. Όχι ότι θα καταψηφίσουμε την έκθεση, απλά δεν θα στηρίξουμε μία σειρά από συμβιβασμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, αλλά ίσως να υποφεληθείτε κύριε εισηγητά τώρα για να μας πείτε όταν θα έχουμε την άτυπη συνάντηση με την Βέλγικη Προεδρία Ποια είναι τα σημεία εκείνα τα οποία ανάλογα με την κατάσταση διαπραγματεύσεων, ποια είναι εκείνα τα σημεία τα οποία για σας θα αποτελούν προτεραιότητα ώστε να τα στηρίξει η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταλαβαίνω ότι έτσι περνάει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια μηνύματα. Οπότε, υποφεληθείτε από την ευκαιρία αυτή για να μας πείτε σε ποια σημεία θέλετε να επιμείνουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους. Θα ξεκινήσω από το τέλος. Ίσως να υπήρξε κάποιο πρόβλημα στην μετάφραση, γιατί εγώ δεν κατάλαβα τελικά ποια είναι τα προβλήματα που έχει η Μαριάν. Εγώ δεν βρήκα καμιά έκφραση που να μην είναι κατανοητή. Πρόκειται για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών όταν πρόκειται για τις αμοιβέ τους από την εργασία. Δυσκολευτήκαμε να βρούμε συμβιβασμό. Οι διάφορες πλευρές έχουν ε, προκαθορισμένες απόψεις. Δημερός πάντως να το συζητήσουμε, γιατί εγώ δεν κατάλαβα ποια είναι αυτή η λέξη που δεν κατάλαβε η συνάδελφος. Όσον αφορά τώρα την ε, Βελγική Προεδρία, θα συναντηθούμε μαζί τους και τόσο το καλύτερο που θα έχουμε αυτή τη συνάντηση πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές, ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί τους πρέπει να δούμε ότι εδώ πρόκειται για μια ειδική περίπτωση συνεργασίας. Το Συμβούλιο πρέπει έτσι καλώς να περιμένει τη γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, όμως το Συμβούλιο μπορεί από την πλευρά του να ακολουθήσει όχι τις απόψεις μας. Ελπίζω να μας ακολουθήσει. Ελπίζω να γίνει αυτό. Ξέρω ότι οι ιδέες μας, οι προτάσεις μας δεν θα γίνουν 100% αποδεκτές από το Συμβούλιο. Όμως, αν μη τι άλλο, ελπίζω κάποια, κάποιες από τις ιδέες μας να τις δεχτεί το Συμβούλιο. Καταφέραμε να συμπεριλάβουμε διάφορες αρχές στο κείμενο αυτό, που εφόσον εγκριθούν από το Συμβούλιο, θα μας καθησυχάσουν. Πρόκειται κυρίως για την προστασία του περιβάλλοντος, για την πλήρη απασχόληση ως τελικό στόχο και πρόκειται βέβαια και για τους επιμέρους στόχους που είπαμε πριν που συμπεριλαμβάνονται στο κείμενο. Και αν θέλουμε νέες θέσεις απασχόλησης πρέπει να επικεντρωνόμαστε στις ομάδες του πληθυσμού που είναι πιο ευάλωτες. Οι νέοι, είπαμε, 15 με 25 ετών, που αποτελούν την κατηγορία ανθρώπων που μπορούν ανα πάσα στιγμή να καλύψουν κάποια θέση απασχόλησης. Αν όμως δεν ενταχθούν έγκαιρα στην αγορά εργασίας, αργότερα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να τους συμπεριλάβουμε. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι είναι σημαντικό να πείσουμε τη Βελγική Προεδρία να ενθαρρύνει τους νέους. Πρέπει και αυτός να είναι ένας επιμέρους στόχος. Οι σοσιαλιστές μας έκαναν κι άλλες προτάσεις. Οι λιγότερο ευνοημένες ομάδες επίσης πρέπει να αποτελέσουν έναν επιμέρου στόχο. Υπάρχουν δηλαδή πολλές δυνατότητες για πολλές ομάδες πληθυσμού. Βάσει αυτού μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ώστε να συμπεριληφθούν περισσότερο τέτοια άτομα στην αγορά εργασίας. Πρέπει να υπάρχει και η καταπολέμηση της φτώχειας στα παιδιά ως επιμέρους στόχος. Γιατί αυτοί που ζουν μέσα στη φτώχεια έχουν πολύ περισσότερες δυσκολίες να μπορέσουν κάποια στιγμή να βρούνε μια δουλειά και να ενταχθούν στην κοινωνία. Δεν υπάρχει αντίφαση ανάμεσα σε αυτή την ιδέα και τη στρατηγική 2020. Υποθέτω ότι αυτές οι ιδέες θα γίνουν αποδεκτές. Αυτές είναι οι για μένα. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, υπογραμμίζουμε την πολιτική συνοχής στην έκθεσή μας. Γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και θα μπορούσαμε ίσως να το βάλουμε όχι στις κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση, αλλά στις κατευθυντήριες γραμμές για την οικονομία ή σε ένα προήμιο ή ανεκτιμώντας κάπου που να μιλάμε για την οικονομία. Εφόσον οι κατευθυντήριε γραμμές για την απασχόληση αποτελούν μέρος της στρατηγικής 2020, η πολιτική συνοχής θα έπρεπε επίσης να αποτελεί ένα τέτοιο σημείο. Πρέπει να υπάρχει συμφωνία μεταξύ των δύο. Αυτά είχα να πω. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την στήριξή σας, αυτό κατάλαβα τουλάχιστον από τα σχόλιά σας. Τώρα αύριο, αν καταφέρουμε να υπερψηφιστούν οι προτάσεις αυτές, τόσο το καλύτερο. Τότε θα συναντηθούμε με τη Βελγική Προεδρία και θα τους το πούμε. Και από εκεί και πέρα είμαι ανοιχτό για συνεργασία με τις διάφορες πολιτικές ομάδες. Μπορούμε να δουλέψουμε ακόμα πάνω στο κείμενο πριν από το Σεπτέμβριο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρή. Αύριο λοιπόν θα ψηφίσουμε την έκθεση αυτή. Και μετά έχουμε τη συνάντηση με την Βελγική Προεδρία. Και το κείμενο θα πάει στην Ολομέλεια για να ψηφιστεί το Σεπτέμβριο. Και μετά το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τις κατευθύνες γραμμές για την απασχόληση, ενώ για την οικονομία έχουν ήδη εγκριθεί. Επόμενο σημείο 5, ανάπτυξη του νομικού θέσεων εργασία στο πλαίσιο μια νέα βιώσιμη οικονομία. Η κυρία Σρέντερ είναι η συγγήτρια. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αύριο λοιπόν θέλουμε να ψηφίσουμε για την έκθεση αυτή και πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων για τη συνεργασία που είχαμε με τους και τις ε, σκιώδεις εισηγητές. Πραγματικά ήταν μια πάρα πολύ παραγωγική διαδικασία η οποία κατά την άποψή μου είχε ο τέλος. Ε, διαπραγματευθήκαμε φόλης της ύλη και τελικά καταλήξαμε σε συμβασμούς. Οι διαπραγματεύσεις άξιζαν τον κόπο Εξάλλου ε, σημειώθηκε επιτυχία γιατί πρόκυψαν ε, και πάρα πολλά κείμενα όπου διορθώθηκαν λάθη. Παραδείγματο χάρη η κυρία Όμεν Ρόιτεν ε, έκανε κάποιες διορθώσεις γιατί κατάλαβε ότι μερικά θέματα δεν ήταν κατανοητά. Κατά την άποψή μου, σε πολιτικό επίπεδο πλησιάσαμε πολύ οι πλευρές ε, μεταξύ τους. Ευχαριστώ λοιπόν τις ε, πολιτικές ομάδες και ευχαριστώ και τις ε, πέντε επιτροπές οι οποίες εμπλούτησαν την έκθεση με τις τροπολογίες τους. Και θα το δείτε αυτό στον κατάλογο ψηφοφορίες. Θα δείτε ότι εγώ συμφωνώ στα περισσότερα πράγματα. Και εκεί που διαφωνώ οφείλεται απλά και μόνο στο ότι προσθέθηκαν άλλα στοιχεία από επιτροπές και όπου λέω ότι ε, παραδείγματος χάνει στην έκθεση Τόμας ε, Μαν υπάρχει αυτό το θέμα της δημογραφίας και δεν πρέπει να το εξετάσω και εγώ. Ε, ήθελα δηλαδή να τραβήξω και κάποιες κόκκινες γραμμές. Υπάρχουν τρεις τροπολογίες από όλες επιτροπές για δημογραφικά θέματα και εκεί και εγώ βάζω την κόκκινη γραμμή και λέω όχι υπάρχει άλλη έκθεση που ασχολείται με αυτό. Αυτά λιγάκι για να καταλάβετε το σκεπτικό. Ή εκεί όπου δηλώνω αποχή κατ' ουσίαν λέω, ναι εντάξει συμφωνώ, αλλά δεν ε, ταιριάζει σε αυτήν την έκθεση ή σε αυτό το σημείο. Ή αναφέρεται στην έκθεση με πολλές λεπτομέρειες. Πάντως ε, θεωρώ ότι όλα αυτά είναι κατανοητά. Ε, πρόκειται για γνωμοδότηση η οποία πρέπει να παραμένει ως τέτοια και μετά να εκφράζονται κάποια στοιχεία με τα οποία συμφωνούμε και εμείς. Γι' αυτό λοιπόν θα ψηφίσουμε, κατ' ουσίαν διαφωνώ, γιατί πρόκειται για ε, επικάλυψη, αλλά δεν είναι θέμα ουσίας. Γι' αυτό λοιπόν σας εξηγώ, γιατί σε ορισμένες τροπολογίες διαφωνώ όπου σας λέω επί της ουσίας συμφωνώ. Δεν είναι λάθος αυτό που λέγεται, μόνο ότι πρόκειται για επικάλυψη. Εκείνο που για μένα είναι το σημαντικότερο είναι εκείνο το οποίο το είπαν τελευταία φορά πολλοί ε, δηλαδή η ανησυχία ότι είναι μια παράλληλη ιστορία με την Ευρώπη 2020. Νομίζω σε όλες τις τροπολογίες καθιστούμε σαφές ότι η στρατηγική διαπραγματεύσεων θα πρέπει να λάβει υπόψη τις αυτές τις εξελίξεις και τα χρηματοδοτικά ε, μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε οι νέες εξελίξεις να ε, προκαλούν την βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό λοιπόν θα ήθελα να υπογραμμίσω κυρίως σε σχέση με το Global Adjustment Fund, με αυτό το ταμείο. Γιατί εκεί προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση. Ε, πολλοί λένε ότι αυτό είναι ένα θέμα ουσίας που δεν πρέπει να επηρεάζει καθόλου τον αρχικό προσανατολισμό του Ταμείου, απλά να πούμε ότι εμείς αναγνωρίζουμε ότι η ε, εξέλιξη της ε, κοινωνίας ε, από τη βιομηχανική κοινωνία στην βιώσιμη ανάπτυξη πράγματι καταργεί αλλά και δημιουργεί θέσεις εργασίας. Νομίζω ότι αυτό ταιριάζει με την έκθεση κυρία Μωρό και επιθυμούμε να κάνουμε να γύρουμε μια γέφυρα προς την έκθεσή της για να μην χαθεί αυτό το στοιχείο. Ελπίζω και θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα ε, ψηφιστεί η έκθεση με μεγάλη ψηφοφορία. Εξάλλου αυτό είπαν οι πολιτικές ομάδες. Όλα τα στοιχεία τα οποία προστέθηκαν από τις ε, πολιτικές ομάδες κατ' ουσίαν ε, λήφθησαν υπόψη στους συμβιβασμούς, στις επιτροπές αλλά και στις δικές μας τις τροπολογίες ακόμα και η διαφοροποίηση ανάμεσα στα διάφορα κοινωνικά μοντέλα νομίζω ότι τώρα είναι σαφέστερη από ό,τι ήταν αρχικά. Ευχαριστώ λοιπόν για τις ε, τροπολογίες που κατατέθηκαν ε, σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας κατόρθωσε να λάβει την απόφαση πριν από το Συμβούλιο. Γνωρίζουμε ότι η Βελγική, όπως είχε συμβεί και με την Ισπανική Προεδρία, ήθελε να βάλει το θέμα αυτό στη μερίσια διάταξη. Εμείς λοιπόν τώρα, αύριο, αν υπερψηφίσουμε την έκθεση, θα έχουμε ε, καταθέσει την πρώτη μας συνεισφορά. Και αυτό ε, θα γίνει ακόμα πιο σαφές όταν Μάλιστα έχουμε τις συζητήσεις με τη Βελγική Προεδρία η οποία έχει αφήσει να νοηθεί ότι θέλει να συμπεριλάβει αυτό το στοιχείο το οποίο εμείς συγκεκριμενοποιήσαμε. Best practice λοιπόν για το πώς εμείς ως Επιτροπή μπορούμε να επηρεάζουμε τις εξελίξεις στο Συμβούλιο. Υπάρχουν κάποιες προφορικές τροπολογίες ε, κάποιες προτάσεις, να βελτιωθεί η διατύπωση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτά μπορούμε να τα δεχτούμε. Βεβαίως ε, για όλες τις ε, προχωρικέ τροπολογίες ε, υπάρχει ένας κανόνας που ισχύει και αυτά έλειψαν υπόψη στη σύνταξη του καταλόγου ψηφοφορίας. Σαφώς εγώ κατά της ε, διαγραφής, αλλά οι περισσότερες ε, διαγραφές ε, αποσύρθηκαν. Υπάρχουν όμως δύο θέματα όπου διαφωνώ. Το ένα είναι ότι θέλω να περιορίσω τα έγγραφα αναφορά σε αυτά που χρησιμοποιεί η Κομισιόν και μόνο. Δεν θέλω να προσθέσω άλλα και εγώ περιορίστηκα, γιατί βεβαίως και εγώ διάβασα πολλά περισσότερα έγγραφα Ίσως θα μπορούσα να τα αναφέρω, αλλά δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα ήταν θετικό. Γι' αυτό λοιπόν περιορίζομαι σε αυτά ε, τα οποία ε, αναφέρει η Κομισιόν ε, ως έγγραφα που τα χρησιμοποίησε. Και αυτό για να παραμένω, παραμείνω στο θέμα. Αυτό το δεύτερο που είναι σημαντικό είναι να παραμείνει ο τίτλος της έκθεσης. Ε, γι' αυτό λοιπόν εγώ είμαι κατά αλλαγής του τίτλου. Αυτά είχα τα σημαντικότερα ήταν αυτά να σας πω. Και τώρα πραγματικά με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ακούσω τι έχουν να παρατηρήσουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Thank Και να ευχαριστήσω την κυρία Σρέντερ, λέει κυρία Σαγιά, για τη δυνατότητα που έχει να κάνει 27 συμβιβασμούς. Νομίζω σωστά το λέω το νούμερο. Πολλές από αυτές θα μπορέσουμε να τις υποστηρίξουμε, όχι όλες βέβαια. Αλλά αυτό που μου αρέσει είναι ότι η βάση αυτής της έκθεσης είναι ο ορισμός του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Βάσει του ορισμού αυτού, όλες οι θέσεις εργασίας μπορούν να γίνουν πιο βιώσιμες, ώστε να μην γίνεται αυτή η διάκριση μεταξύ καλής και κακής βιομηχανίας. Όλες οι θέσεις εργασίας μπορεί να είναι πιο βιώσιμες. Αυτό λοιπόν είναι η βάση της έκθεσης και η πολιτική μας ομάδα θα ήθελε βέβαια να μην υπάρχει αυτός ο όρος ε, green, πράσινος, και να μιλάμε για βιώσιμες θέσεις εργασίας και όχι για πράσινες θέσεις εργασίας. Και οι περισσότερες από τις προφορικές τροπολογίες που θα καταθέσουμε είναι για να αλλάξουν αυτοί οι ορισμοί για τις πράσινες θέσεις εργασίας. Όπως σας είπα στις διαπραγματεύσεις μας, δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούμε τις δυνατότητες θέσεων εργασίας που μας προσφέρουν αυτές οι νέες ε, δυνατότητες για πιο βιώσιμες θέσεις εργασίας, να τις λαμβάνουμε υπόψη, αλλά να μην είμαστε υπεραισιόδοξοι. Ε, η ελπίδα ότι μπορεί να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται και από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες χάνονται ακριβώς επειδή αλλάζει τεχνολογία. Και νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ο ρεαλισμός άλλωστε είναι η βάση του ΕΛΚ. Υπάρχουν τώρα κάποια θέματα στους συμβιβασμούς. Παραδείγματος χάρη στο συμβιβασμό BB, που θα έχει δεσμευτικούς στόχους και κυρώσεις για τα κράτη-μέλη που δεν έχουν καλή απόδοση. Νομίζω ότι εδώ υπερβαίνουμε τα σκαμμένα και ε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε αυτό το συμβασμό. Στο συμβασμό G Having uh, also binding conditions. Και πάλι υπάρχουν δεσμεύσεις για τουλάχιστον 10 χρόνια, λέει ο συμβασμός, με τις αλλαγές όμως της τεχνολογίας νομίζω ότι τα 10 χρόνια είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Εάν υπάρχουν επιδοτήσεις ή φορολογικές ελαφρύνσεις για 10 χρόνια, ίσως να είναι κατασπατάληση χρημάτων αυτό. Πλέον είναι τόσο ταχύες οι αλλαγές στη τεχνολογία που θα πρέπει να το λαμβάνουμε και αυτό υπόψη η συγγήτρια αναφέρθηκε στην παράγραφο 19 και εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο προβληματική αυτή η παράγραφος. Εγώ πραγματικά ελπίζω να μπορέσει να αλλάξει ο στόχο του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και αν μπορέσουμε να το διευκρινίσουμε αυτό λίγο περαιτέρω στο τέλος θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για μας. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ε, είναι οι πιο σημαντικέ παρατηρήσει μου. Αν τι κατάλαβε κανεί, ο Τόμα και η κυρία Χάρκιν στη συνέχεια. Συνήθω ε, ήθιστε να λέμε ευχαριστούμε την εισηγήτρια. Ξέρετε, αυτή τη φορά πραγματικά το εννοούμε. Ε, γιατί είδαμε Ελιζαμπέτ ε, τη δύναμη με την οποία δούλεψες ε, και εγώ θέλησα να συγκεράσουμε τις ε, αντικρουόμενες απόψεις, εσύ τα κατάφερες μια χαρά, κάναμε πάρα πολλές συζητήσεις και στόχος μας ήταν να δούμε πώς μπορούμε να συμπεριλάβουμε και διαφορετικές θέσεις. Άρα δηλαδή ε, πρέπει να ικανοποιηθούμε ή σκεφτόμαστε να ικανοποιηθούμε με μια διατύπωση που μόλις θα πετύχει την πλειοψηφία ή να αναζητήσουμε ε, κάτι παραπάνω. Πράγματι υπάρχουν κάποιες επικαλύψεις που είναι περιττές, εντάξει, θα το λάβουμε αυτό υπόψη μας γιατί μερικές φορές ξέρετε κάτι, γράφει κανείς μια εκθέση και μετά έρχονται τόσες ε, προσθήκες που αναγκάζεται κανείς να κάνει και πολλές αλλαγές. Δεν συνέβη όμως αυτό. Ούτε εγώ θέλω να έχουμε επικαλύψεις. Δεν θέλω θέματα που εμφανίζονται σε άλλες εκθέσεις να εμφανίζονται και εδώ. Γιατί στο τέλος ε, θα έχουμε ε, μορφώματα υπερβολικά, αντιπαθητικά που δεν μ' αρέσει. Ε, και αυτό που έχει σημασία είναι πώς μπορεί κανείς να επιτύχει ευρωπαϊκή υπεραξία. Ίσως μπορούμε να πούμε στους ε, δημοσιογράφους και να τους δείξουμε πώς είναι δυνατόν Αποτελεί τελείως διαφορετικές θέσεις να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να ικανοποιεί όλου. Αυτό είναι ένα θέμα που αξίζει τον κόπο να το εξετάσει κανείς και πέρα από αυτήν την έκθεση γιατί μερικοί ε, έξω οι πολίτες πιστεύουν ότι απλά ε, με κάποια ισχνή πλειοψηφία περνάνε εκθέσεις. Δεν είναι αλήθεια. Βλέπουμε ότι διαμορφώνονται και ουσιαστικές πλειοψηφίες και βλέπουμε επίσης ότι η έκθεση αυτή άξιζε τον κόπο. Τι πνεύμα συνεργασία είναι αυτό που επικρατεί εδώ στην Επιτροπή μα, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Χάρκιν. Ε, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια εκ μέρου του κυρίου Στέρξ που είναι σκιώδη ηγητή και είναι σε κάποια άλλη επιτροπή αυτή τη στιγμή. Καταρχά, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Σρέντερ για τι συμβιβαστικέ ε, τροπολογίε, διότι έλαβε υπόψη τι απόψει των άλλων Ευρωβουλευτών και τι έλαβε υπό... τις συμπεριέλαβε και γι' αυτό λοιπόν δέχεται τι περισσότερε. Επίση, θα ήθελα να αποσύρει κάποιε από τι τροπολογίε που ζητούν διαγραφή, διότι άλλαξαν με τέτοιο τρόπο οι παράγραφοι για τι οποίε δεν έχει πρόβλημα και νομίζω ότι αυτά το έχει συζητήσει με την κυρία Σρέντερ. Ο συμβιβασμό BB είναι αυτό ο οποίο δεν μπορεί να δεχτεί, διότι αναφέρεται στου δεσμευτικού στόχου, κάποιο το είπε αυτό πριν, και επίση επικρίνει τη στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, μια στρατηγική την οποία έχουμε συμφωνήσει με όλοι και μάλιστα πέρασε και σχετικό κείμενο στο Κοινοβούλιο πρόσφατα. Θα ήθελα να κάνω και δύο σχόλια προσωπικά. Μόλι διάβασα το τελικό σχέδιο κειμένου των συμβαστικών τροπολογιών, να συγχαρώ την κυρία Σρέντερ Πρόκειται για μια έκθεση η οποία θεωρώ ότι είναι πολύ στοχευμένη και πολύ συνεκτική και εξαιρετική φυσικά, αλλά αυτό είναι αυτονόητο. Και τέλος, θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την παράγραφο 19 και πάλι, για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Εδώ στοχεύουμε στον εργαζομένο και, στον στις απαιτήσει του και αν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη οικονομία, θα μπορούσαμε να έχουμε μια περίπτωση στην οποία μπορεί κάποιος εργαζόμενος να αποφασίσει να έχει μια τοπική ε, επιχείρηση μεταφορών ε, στην Ήπεθρο και αυτό μπορεί να μην θεωρείται βιώσιμο. Δεν θα ήθελα να περιορίσουμε το ε, πεδίο εφαρμογή του Ταμείου Προσαρμογή στην Παγκοσμιοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Η Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Μετά από αυτά που είπε η Μαρία Ναρκίν, ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Σρέντερ, που όντως με πνεύμα συνεργασίας ετοίμασε την εκθεσή της. Προσφέρει πολλά η εκθέση αυτή, αλλά για το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, η κυρία Σρέντερ προσπάθησε να οργανώσει την έκθεσή της με τέτοιο τρόπο που είναι την ίδια γραμμή με την έκθεση που κάνουμε. Και όπως είπε και η Μαρία Χάρκιν, δεν μπορούμε να περιορίσουμε το στόχο εδώ μόνο για το Ταμείο Προσαρμογή του Παγκοσμιοποίηση. Δεν μπορούμε να το περιορίσουμε μόνο στην αηφόρα ανάπτυξη. Υπάρχει σε άλλες τροπολογίες και προτιμάω κατά πολύ την τροπολογία του κύριου Πουπάκη και της κυρίας Γκρούνη για την μελλοντική απασχόληση. Δηλαδή, όποιος και αν είναι ο τομέας, το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση έχει φτιαχτεί για να προετοιμάσει τους μισθωτούς να γράφονται σε μία βιώσιμη δραστηριότητα που θα κρατήσει στο μέλλον και όχι προσωρινή. Το είπε η κυρία Χάρκιν. Τώρα, εφόσον με επιτρέπετε κυρία Πρόεδρε, στο κείμενο της έκθεσης πρέπει να αλλάξουμε μια λέξη, γιατί ίσως να παρασυρθήκαμε. Σελίδα 13-13. Γίνεται μνήα στην Ανατολική Γερμανία. Λέει αυτοί που δουλεύουν από την Ανατολική Γερμανία κτλ. Ε, Γερμανία φτάνει νομίζω γιατί εδώ και χρόνια δεν έχουμε πια άλλη Γερμανία, έχουμε μία ενωπημένη Γερμανία. Συνεπώς αυτό το ανατολική μπορεί να βγει. Γιατί είναι για τα αρχεία μας μόνο και τίποτα άλλο. Ιστορικός όρος και όχι σύγχρονος. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ό,τι θέλετε, αλλά η συγγήτρια θα κρίνει αν συμφωνεί με αυτήν την ιστορική διόρθωση όχι. Αλλά ίσως να είναι και θέμα μετάφρασης, ε. Ίσως να αναφέρονταν στις ανατολικές περιοχές της Γερμανίας. Δεν ξέρω, πρέπει να το δούμε. Στα γαλλικά μπορεί να υπάρχει πρόβλημα όντως. Η κυρία Γκρούνη και μετά ο κύριος Λουμπίτσον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ την κυρία Σρέντερ πρώτα απ' όλα για τις τροπολογίες της και τις συμβαστικές και για όλη της τη δουλειά. Είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για τις αυριανές θέσεις απασχόλησης. Εγώ συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε εδώ πριν, αλλά έχω να προσθέσω κάτι. Είχα υποβάλει μια τροπολογία για τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου για τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος. Δεν ε, εγκρίθηκε και μου εξηγήσανε για ποιο λόγο. Βρέθηκε ένας συμβιβασμό για να γίνει μια μελέτη σκοπιμότητας για αυτές τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος. Όμως υπάρχει και κάτι που πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε. Στην επιχείρηση πάντα φτάνουμε με καθυστέρηση όσον αφορά την εκπαίδευση, την κατάρτιση. Και κατόπιν ορτής διαπιστώνουμε ότι έχουμε ανθρώπους που βρίσκονται στην ανεργία και από την άλλη μεριά επιχειρήσεις που ψάχνουν προσωπικό. Αφού λοιπόν κάνουμε έρευνες σε ένα σωρό πράγματα, δεν θα έπρεπε να είμαστε σε θέση να δούμε περισσότερο μακροπρόθεσμα και καλύτερα, ώστε να ξέρουμε τι ε, απασχόληση θα χρειάζεται. Για τον ηλιακό τομέα αναφέρουμε εδώ πριν δεν υπήρχαν τέτοιες θέσεις απασχόλησης. Όταν ήμουν εγώ φοιτήτρια δεν μιλούσαμε καν για την ποιότητα των επιχειρήσεων. Ενώ σήμερα υπάρχουν ε, ανάγκες για τέτοιες θέσεις απασχόλησης. Με δύο λόγια, η κατάρτιση που γίνεται για να προετοιμάσουμε τους νέους για την απασχόληση δεν ασχολείται αρκετά με το μέλλον. Ούτε η δημόσια εκπαίδευση ασχολείται με αυτό, το κράτος. Γι' αυτό θα έπρεπε να το σκεφτούμε περισσότερο και από ευρωπαϊκό επίπεδο να βοηθήσουμε σε αυτόν τον προβληματισμό για να είναι έτοιμος ο κόσμος για τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος. Ευχαριστούμε, λέει ο κύριος Λουίξον. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, κυρία Σρούντερ και τους ε, άλλους συναδέλφους για την πολύ καλή συνεργασία. Πιστεύω λοιπόν ότι παρότι για αυτές ε, τις ε, τροπολογίες υπήρξε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τελικά καταλήξαμε σε συμβασμούς ε, τους οποίους οι περισσότεροι από εμάς θα τους δεχθούμε. Θα έχουμε να κάνουμε με μια ιδιαίτερα ισόρροπη έκθεση που λαμβάνει όλα τα κριτήρια υπόψη που είναι απαραίτητα για να επιτύχουμε αυτή την αλλαγή που επιθυμούμε. Με πολύ μεγάλη χαρά διαπιστώνω ότι ιδιαίτερα η εκπαίδευση, η έρευνα, οι ίσες ευκαιρίες και κυρίως ε, το πρόβλημα της ανεργίας των νέων. Αυτά τα θέματα προβάλλονται στην έκθεση και ας μην ξεχνάμε ότι σε περίοδους ε, κρίσης η πολιτική απασχόληση είναι πολύ μεγάλη σημασίας. Οι νέοι οι άνδρες και οι γυναίκες πρέπει όλοι να συμβάλλουν στο να αλλάξει η κατάσταση. Παράλληλα όμως δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι με μονομένη τομή σε λόγω ιδιαίτερων μέτρων ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προβλήματα. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω να έχει ζητήσει κανένα άλλο το λόγο, οπότε η συγκήτρια. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ σκέφτηκα κατά πόσον ε, σε αυτό το Global Adjustment Fund θα μπορούμε να καταλήξουμε ε, σε κάποια λύση, γιατί νομίζω ότι κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα της κατανόησης. Είναι δηλαδή το εξής. Εγώ πίστευα ότι πρέπει να αλλάξει τελείω. Όμως ε, τελικά νομίζω θα βρούμε κάποια λύση και θα προσπαθήσω να το δούμε πολύ προσεκτικά. Εσείς θέλετε τα χρήματα να μπορεί κανείς να τα ε, χρησιμοποιήσει εφόσον προσφέρονται. Αυτό βέβαια αλλάζει την κατάσταση, γιατί ε, και η κατάσταση επιτόπου μπορεί να αλλάξει. Τέλος πάντων το κατάλαβα, θα το ξαναδώ. Ε, είδα λιγάκι τώρα τις διατυπώσεις και ίσως μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, έτσι ώστε να μην είσαστε αναγκασμένοι να είσαστε κατά των πάντων. Θα το δούμε λοιπόν. Κυρία Σάια, γιατί δεν θέλω να συμπεριλάβω τη δική σας τη διατύπωση με bad και good interest. Ακριβώς με το λόγο που θέλετε εσείς να προσθεθεί. Εγώ δεν θέλω η βιομηχανία να είναι καλή ή κακή και γι' αυτό δεν θέλω αυτή τη διατύπωση. Εσείς ε, θέλετε αυτή τη διατύπωση, εγώ διαφωνώ διότι την κλασική βιομηχανία τη χρειαζόμαστε. Ε, χωρίς τη χαλιβουργία, ε, ας είμαστε ειλικρινεί, ε, δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τους ανεμόμυλους. Γι' αυτό λοιπόν είμαι κατά της δικής σας διατύπωση. Εσείς μιλάτε για το καλό κακός, good bad industry και εγώ δεν συμφωνώ. Αυτό είναι ο λόγος. Τελικά νομίζω συμφωνούμε και αν καταλάβετε κι εσείς ότι η δική μου διατύπωση είναι τέτοια που δεν οδηγεί στο να γίνεται αυτή η διαφοροποίηση καλής ή κακής βιομηχανίας, δεν χρειάζεται και να το τονίζουμε. Η συμβαστική ε, πρόταση του κυρίου Μαν λέει ότι ε, έχουμε αλλαγές σε όλους τους ε, βιομηχανικούς κλάδους, αυτό έχει επιπτώσεις θέσεις εργασίας και το καθεξής. Και από όλα αυτά ε, προκύπτει και το ερώτημα που έθιξε η κυρία Κούνη. Δηλαδή οι έρευνες κατέδειξαν ότι δεν υπάρχουν αυτές οι νέες θέσεις εργασίας με το νέο προφίλ. Έχουμε παραδοσιακά επαγγέλματα, ε, μεταποιητικά επαγγέλματα που εγκυμονούν νέα στοιχεία. Δηλαδή, ο υδραυλικός μπορεί να είναι 15 ετών και να είναι τέλειος και τις δικές του τις ικανότητες τις χρειάζομαι για να μπορέσω να εγκαταστήσω ένα θαυμάσιο ηλιακό θερμοσύφωνα. Αυτός λοιπόν πρέπει να βελτιώσει τις γνώσεις του και να μάθει πώς μπορεί να συνδυάσει τον ηλιακό με τον ηλεκτρικό θερμοσύφωνα. Εγώ λοιπόν πρέπει να του δώσω αυτή τη δυνατότητα της ε, περαιτέρω εκπαίδευσης ε, για να μπορεί και αυτός να εργαστεί. Ξέρετε, έχουμε τεράστια έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, κυρίως υδραυλικών. Κυρία Μωρό, εσείς ρωτήσατε... Ε, γιατί ακριβώ έγραψα το παρόμοιο στη δήλωση. Α πω ένα παράδειγμα. Στη Γερμανία, ή αναφέρθηκα γιατί αναφέρθηκα στην Ανατολική Γερμανία. Στη Γερμανία, ξέρετε, ε, τα κέντρα ηλιακή ενέργεια ε, είναι κυρίω στην πρώην Ανατολική, είναι 4-5. Ε, και γι' αυτό αναφέρω αυτό το παράδειγμα. Είναι καθαρά γεωγραφική η περιγραφή θα μπορούσα να αναφέρω τα διάφορα κρατήδια, αλλά εδώ είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι μια περιοχή στη Γερμανία που ήταν ιδιαίτερα μειονεκτική με αυτά τα νέα κλάστερ, ε, αυτές τις ομάδες, τα γκρουπ ε, βιομηχανικών μονάδων, έχει σημειώσει μεγάλη πρόοδο γιατί σα επαναλαμβάνω, ήταν η πιο μενεκτική περιοχή στη Γερμανία. Έχει έμεσα σχέση με την ιστορία, απλά ο όρος που χρησιμοποιώ εγώ είναι καθαρά γεωγραφικό. Γι' αυτό σα το εξηγώ, δεν έχει νόημα τώρα εδώ να το αλλάξουμε, Σα εξηγώ τι εννοώ. Τα 10 χρόνια, γιατί αναφέρω τα 10 χρόνια, διότι το... Ευρώπη 2020 θα είναι μετά από 10 χρόνια. Γι' αυτό μιλάμε και για το διάστημα των 10 ετών. Τώρα μιλάμε για στρατηγικές στο πλαίσιο της ε, Ευρώπης 2020 για ένα δεκαετές διάστημα. Είναι λοιπόν ένα διάστημα που ταιριάζει για να δημιουργηθούν οι συνθήκες πλαίσιο. Αυτό κάνουμε με τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης ή με τη στρατηγική του κυρίου Μπαρόζο. Αυτό είναι ο λόγος που αναφέρουμε το διάστημα των δεκατών. Μπορούμε να μιλήσουμε και για 20 χρόνια. Δεν έχει όμως νόημα. Θέλουμε να έχουμε ακριβώς αυτό το συνδυασμό ε, με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Δεν θέλουμε να έχουμε κάτι ξεχωριστό θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να γράψει σε παρένθεση ακριβώς όπως αναφέρεται στη στρατηγική 2020, αλλά αυτό και πάλι θα αποκαλούσε ε, πλατιασμό στην έκθεση. Νομίζω ότι είπα τα σημαντικότερα. Α, και κάτι άλλο. Πολλοί εκφράστηκαν κατά της ε, τροπολογίας BB. Αυτό ε, δεν το είπα μόνο εγώ, προέκυψε και από τροπολογίες αυτής της Επιτροπής. Εγώ το μόνο που έκανα ήταν να προσπαθήσω με τις τροπολογίες να βρω μια διατύπωση που δεν θα περιλαμβάνει επαναλήψεις. Οι συνάδελφοι όμως έκαναν την πρόταση, εγώ θεωρώ ότι είναι καλή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και μία πρόταση από την Επιτροπή, όχι από εμένα. Και γι' αυτό ε, νομίζω πρέπει να στηριχθεί αυτή η τροπολογία και θελήσαμε απλά να βελτιώσουμε τη διατύπωση. Γι' αυτό λοιπόν ε, βρήκαμε με τον συντάκτη των τροπολογιών αυτή τη διατύπωση. Αυτή είναι η τροπολογία BB, είναι πολιτικής φύσης, εγώ τη στηρίζω και ελπίζω να βρεθούν και κάποιοι συνάδελφοι που να με στηρίξουν. Παναλαμβάνω, δεν την ανακάλυψα εγώ την τροπολογία. Ήρθε από την Επιτροπή. Και ο συντάκτης της ε, τροπολογίας είπε ότι μόνο με τον τρόπο αυτό μπορώ να επιτύχω το στόχο μου. Ε, και δεν μπορώ και εγώ να του πω, δεν ε, θέλω ούτε να το ακούσω. Εγώ αναγνωρίζω την εμπειρία του συντάκτη αυτής της τροπολογίας. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κυρία Μωράν. Στα αγγλικά μιλάει για Eastern Germany. Οπότε είναι θέμα μετάφρασης του εκτιμώντας του συγκεκριμένου. Δεν ξέρω πώς διορθώνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αύριο θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Σρέντερ και θα πάει το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Τώρα ερχόμαστε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης. Είναι η γνωμοδότηση του συναδέρφου μας Τόμας Μαν, λέει η πρόεδρος, για τις γυναίκες εργαζόμενες σε επισφελείς θέσεις απασχόλησης. Τόμας Μαν είπα, πω πολύ πρόεδρος, είδατε από το πολύ πνεύμα συνεργασίας που έχουμε εδώ στην Επιτροπή μας, τα μπλεξα. Λάθος έκανα, λάθος. Τόμας Χέντελ, συγγνώμη. Συγγνώμη ζητώ από τον εισηγητή, λέει πρόεδρος. Είναι γνωμοδότηση που πάει στην Επιτροπή για τα Δικαιώματα της Γυναίκας. Έχετε το λόγο κύριε εισηγητά. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αν ο κύριος Τόμας Μάν θέλει να πάρει την έκθεσή μου, με πολύ μεγάλη μου χαρά. Και εγώ θα τη ε, συζητήσω, θα τοποθετηθώ επ' αυτή, θα είναι πολύ ενδιαφέρον νομίζω το όλο θέμα και η εξέλιξη. Η γνωμοδότηση που σας ε, κατέθεσα δεν είναι ότι χρειάζεται να την εξηγήσω ιδιαίτερα. Ε, κυρίως ε, οι γυναίκες τα τελευταία χρόνια έχουν εξωθηθεί σε επισφαλείς θέσεις εργασίας. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στην Ευρώπη αλλά και ανά τον κόσμο υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά την ποιότητα της εργασίας, τις αμοιβέ, αλλά και τις ευκαιρίες να βρει κανεί απασχόληση. Γι' αυτό λοιπόν η Επιτροπή μας ε, πρέπει να συμφωνήσει ε, με αυτά που λέει η Επιτροπή Γυναικών και να τους ε, δώσουμε και μία γνωμοδότηση. Εγώ ευθύ εξ αρχής ευχαριστώ όσους κατέθεσαν τροπολογίες. Είναι μάλιστα πάρα πολλές αυτές. Και αυτές συνέβαλαν στο να διευρύνω τη γνωμοδότησή μου, να τη συμπληρώσω με πολλούς δεύτερους υποστόχους. Εγώ λοιπόν ε, είμαι ευγνώμων σε όσους κατέθεσαν τροπολογίες γιατί ακριβώ ανέφεραν πάρα πολλές και προσέθεσαν πάρα πολλές αποχρώσεις. Εγώ ε, συστήνω πολλές από αυτές τις ε, αποχρώσεις να τις εγκρίνουμε. Μόνο κάποιες από τις τροπολογίες θα τις συστήνω να τις καταψηφίσουμε. Κυρίως θα αναφέρω ένα θέμα Πρόκειται για το θέμα του ε, κατώτατου μισθού. Αυτή η διατύπωση περί κατώτατου μισθού ε, δεν έγινε αποδεκτή από όλους. Και θέλω να σε επισημάνω ότι εδώ δεν πρόκειται για μία οδηγία, πρόκειται για κατανόηση, για συμφωνία πάνω σε ένα στόχο. Δηλαδή με ποιο τρόπο θα εφαρμοστούν αυτά από τα κράτη-μέλη. Αυτό βέβαια είναι ε, δική τους υπόθεση των κρατών μελών. Κατά πόσον θα εφαρμόζουν το το μισθό τομεακά, περιφερειακά ή εθνικά, αυτό είναι θέμα των κρατών μελών. Και αναφέρομαι κυρίως ε, στους συναδέλφους από τις νότιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζω τις επιφυλάξεις τους. Δεν πρόκειται εδώ για μια ενιαία ρύθμιση στην Ευρώπη έτσι ώστε να αντικατασταθούν οι διατάξεις περί κατώτατου μισθού. Κάθε άλλο. Δεν εννοούμε αυτό η διατύπωση αυτή η οποία αύριο θα σας ε, κατατεθεί με τη μορφή συμβαστικής ε, τροπολογίας αυτή η διατύπωση ε, ταιριάζει σε όλες τις, τις, τους εθνικούς κανονισμούς. Έχουμε σε 21 χώρες από τις 27 όπου υπάρχουν ρυθμίσεις περί κατώτατου μισθού. Όμως θα πρέπει να συμφωνήσουμε πάνω σε ένα στόχο που δεν είναι νέος στο Κοινοβούλιο, δηλαδή να εξευρεθεί ένας κατώτατος μισθός που να είναι το 60% του εκάστοτε εθνικού μέσου μισθού. Τώρα, ε, κατά πόσον αυτό μπορεί να εφαρμοστεί, όπως σας είπα, αυτό δεν είναι θέμα της οδηγίας, αυτό είναι θέμα ενός πλαισίου και στόχων πάνω ε, στους οποίους πρέπει κανείς να συμφωνήσει. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε συνδυασμό με τις ε, συμβαστικές προτάσεις. Στην έκθεση αυτή θίγουμε και το θέμα της ίσης αμοιβή για την ίδια εργασία. Εγώ ελπίζω ότι αύριο πολλοί από τους συναδέλφους θα συμφωνήσουν με αυτή τη γνωμοδότηση. Στην Επιτροπή για την Ισότητα των Δύο Φύλων, αυτά που είπαμε ε, έγιναν ευρέως αποδεκτά και ελπίζω λοιπόν ότι αύριο για αυτόν τον λόγο θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε την έκθεσή μου αυτή, τη γνωμοδότηση. Κυρία Βάσιο, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Τόμας Χάντελ για τις καλέ του συστάσεις και για την έκθεσή του. Δεν είμαστε βέβαια επί τη ουσία αρμόδια επιτροπή. Το πρόβλημα των συμβολέων αυτών επισφαλούς εργασίας ε, είναι κάτι που έχει επιδεινωθεί, ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση που γίνεται όλο και περισσότερο κοινωνική κρίση. Θα μπορούσα να αναφερθώ σε διάφορες χώρες της, ε, της Ευρώπης. Η Βουλγαρία έχει ξεχαστεί κάπως. Εκεί έχουμε ξεχάσει τα συμβόλαια αυτά ή κάποια εποχή τα είχαμε ξεχάσει επειδή η κατάσταση είχε βελτιωθεί κατασταση εχει Όμως τώρα με την οικονομική κρίση οι γυναίκες όλο και περισσότερο φοβούνται να δηλώσουν ότι έχουν τέτοια συμβόλαια επισφαλούς εργασίας, ότι δεν έχουν δικαιώματα για άδεια για ασφάλιση κλπ. κλπ. Με δύο λόγια φοβούνται να πούν ότι δουλεύουν στις επιχειρήσεις που δίνουν τέτοια συμβόλαια και κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύουν. Γι' αυτό θα έπρεπε, πιστεύω, να βρούμε έναν τρόπο η έκθεση αυτή να γίνει γνωστή στην κοινή γνώμη της Ευρώπης. Γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι αναγκάζονται να δουλέψουν κάτω από τέτοιες επισφαλείς συνθήκες εργασίας και εφόσον γίνει γνωστή η έκθεση αυτή σε αυτούς θα νιώσουν ότι έχουν ένα σύμμαχο μαζί τους, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή. Εδώ και καιρό επιμένουμε για το ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή ε, νομοθετούν για τους ε, εποχιακούς εργαζόμενους. Για πολλούς συναδέρφους, όρος αυτός, εποχιακοί εργαζόμενοι, έτσι όπως είναι γνωστό στην Ανατολική Ευρώπη ή έτσι όπως εφαρμόζεται στην Νότια Ευρώπη, είναι κάτι άλλο. Πρόκειται για εποχιακούς εργαζόμενους που δουλεύουν στη Γεωργία, που δουλεύουν ε, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα κάτω από συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα συμβόλαια που έχουν είναι παράνομα, πληρώνονται σε ρευστό χωρίς να έχουν καμία απολύτως κοινωνική προστασία. Θέλω επίσης να αναφερθώ λίγο και στο θέμα που έθεσε και ο κύριος Έντελ. Δηλαδή 60% του κατώτατου, μάλλον του μέσου μισθού, 60% του μέσου μισθού να είναι ο κατώτατος μισθός, είναι κάτι που έχει δημιουργήσει μια μεγάλη συζήτηση δεν είναι θέμα γλωσσικό. Πρόκειται για έσοδα, πρόκειται για μισθό. Οι όροι σημαίνουν διαφορετικά πράγματα στις διάφορες γλώσσες. Ένα μεγάλο μέρος των συναδέλφων ήταν κατά του κειμένου, όχι μόνο γιατί πιστεύουν ότι δεν υπάρχει όρος κατώτατος μισθός σε πολλές χώρες, αλλά και επειδή είναι συλλογικέ συμβάσει τα συνδικάτα οι κυβερνήσει που αποφασίζουν για αυτόν τον κατώτατο μισθό. Αλλά επίση επειδή πολλοί συνάδελφοι πιστεύουν ότι πρόκειται για μια πολιτική που έχει να κάνει με την επικουρικότητα και όχι με την κοινοτική πολιτική. Οι σοσιαλδημοκράτες δεν θα υποστηρίξουν αυτόν τον συμβιβασμό. Πάντως θα περιμένουμε και την τελική έκδοση του κειμένου για να δούμε. Η κυρία Τσιν Λάπερ και η κυρία Μαριάν Χάνκερ. Η κυρία Λάμπερτ πρώτα. thank you. Ευχαριστώ. Φαίνεται να δημιουργούνται δυσκολίες εδώ. Αν μιλάμε για διαφορές μεταξύ εισοδήματος και μισθού, νομίζω ότι είναι σαφές ότι ο μισθός είναι αυτό το οποίο ε, λαμβάνει για αυτό που έκανε. Και αυτό δεν είναι απαραίτητο το ίδιο με το εισόδημα που μπορεί να είναι από την περιουσία σου, από το καταπίστευμά σου ή από ε, επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης. Ε, ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έθεσε και η κυρία Χάρκιν στη συνεδρία των συντονιστών την περασμένη εβδομάδα. Να δούμε δηλαδή εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κατάλληλη ορολογία και να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούμε. Στο, συμβιβαστικό, στο συμβιβασμό C αυτό αναφέρουμε, αυτό το οποίο λαμβάνεις για το έργο που προσφέρεις. Και όπως είπαμε, αυτό βρίσκεται σε όλα τα θέματα που άπτονται επίπεδων φτώχειας, αλλά μιλάμε για αυτό το επίπεδο που αναφέρει ο συμβιβασμό. Ε, το να βρίσκεται κάποιος ε, στο επίπεδο της φτώχειας ή στον κίνδυνο της φτώχειας και αν κάποιος ε, βρίσκεται σε πληρωμένη εργασία θα πρέπει να αναφέρεται αυτό το οποίο λαμβάνει. Δεν νομίζω ότι είναι επαναστατικό αυτό. Υπάρχουν και διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει και ε, ο τρόπος με τον οποίο μπορείς να επιτύχεις το στόχο είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Δεν λέμε ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν αυτό ή αυτό είναι το ποσό το οποίο θα πρέπει να καθορίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ε, ελάχιστος μισθός σε όλη την Ευρώπη. Δράτω με δε τις ευκαιρίες επειδή έχω το λόγο να πω ότι με εκπλήσει το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια ε, με τόσες οδηγίες για θέματα ισότητας των φύλων ακόμα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ισότιμος μισθός ε, για ισότιμη εργασία. Με εκπλήσει το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια δεν το έχουμε επιτύχει όσον αφορά στους εποχιακούς εργαζόμενους Έχω την αίσθηση ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρότασή της για τους εποχικά εργαζόμενου, το οποίο θα το συζητήσει σίγουρα η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, αλλά σίγουρα και η Επιτροπή μας, διότι αναφέρεται και στα δικαιώματα και όχι μόνο ε, στην, ε, στα προβλήματα αυτά. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Χέντελ για την εξαιρετική του δουλειά και την αγαστή συνεργασία που είχαμε στο θέμα αυτό. Κάποια σύντομα σχόλια ε, για τους συμβιβασμούς. Ο συμβιβασμός Α μας δημιουργεί πρόβλημα στην ενότητα που αναφέρεται, ενθαρρύνει την ανάγκη κλπ. κλπ. Θα έπρεπε να λέμε επισημένη, notes, συνήθως λέμε τονίζει, στρέσες, το αλλάξαμε για να είναι πιο αποτελεκτό... αλλά το ενθαρρύνει δεν είναι και πολύ λογικό, τουλάχιστον στα αγγλικά. Δεν ξέρω πώς είναι στις άλλες γλωσσικές εκδοχές. Επίσης, μας ενδιαφέρει το θέμα της πρόσβασης σε πλήρη κοινωνική ασφάλεια, ασφάλιση, όταν κάποιος ε, απασχολείται όχι με πλήρη απασχόληση. Ε, σε κάποιες χώρες υπάρχει θέμα με το, ε, την κοινωνική ασφάλιση που λαμβάνεται. Αν διαγράψουμε τον όρο πλήρης ε, κοινωνική ασφάλιση, ε, ίσως να μπορέσουμε να βρούμε κάτι. Μπορεί να ζητήσουμε κατά τμήματα πληροφο, ε, ψηφοφορία. Θα το συζητήσουμε με το συντάκτη της γνωμοδότησης. Ο συμβιβασμός εσύ μας δημιουργεί πρόβλημα. Το ανέφεραν και άλλοι εδώ. Δεν θα επισέλθω σε λεπτομέρειες, ε, τα επιχειρήματα τα ακούσαμε, αλλά έχουμε πρόβλημα με το συμβιβασμό αυτό. Οι άλλοι συμβιβασμοί είναι καλοί, αλλά η προφορική τροπολογία εδώ δεν ξέρω, η τροπολογία που ε, έχω εγώ, η προφορική, στην παράγραφο 8, διαφέρει από την τροπολογία που έχουμε στον κατάλογο ψηφοφοριών και λέει καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην οδηγία για την απόσπαση εργαζομένων του τομεί τη υγεία, τη μέρημνα, των ξενοδοχείων και τη γαστρονομία, καθώ και τη κατοίκων υπηρεσία στην απόσπαση των εργαζομένων. Στον κατάλογο των ψηφοφοριών δεν περιλαμβάνεται η φράση αυτή. Εάν υπάρχει αυτή η φράση, Ούτως ή άλλως, εξετάζουμε το θέμα της αναθεώρησης ε, της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων. Δεν είμαι βέβαιη ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί, να, μπορεί κάποιος να μου το διευκρινίσει. Δεν είμαι βέβαιη ότι μπορούμε να συμπεριλάβουμε τους εργαζόμενους του τομείς της υγείας. Θα πρέπει να εξετάσουμε το θέμα των άλλων κατηγοριών εργαζομένων. Θα πρέπει να το δούμε στο θέμα της αναθεώρησης. Ίσως μπορεί να μου το εξηγήσει και ο συντάκτης της γνωμοδότησης αν το σωστό δηλαδή είναι αυτό που έχω στον κατάλογο ψηφοφοριών ή τον κατάλογο που έχω με την προφορική τροπολογία. Ο κύριος Κρίστενσεν και μετά ο κύριος Τόμας Μάν. Θα ήθελα να σας εξηγήσω πολύ σύντομα γιατί εμείς από πλευράς βορείων χωρών έχουμε κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά αυτή την έννοια του κατώτατου μισθού ή αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο ορίζεται ο κατώτατος μισθός. Γιατί όταν γίνεται ένας τέτοιος υπολογισμός, κατ' ουσία επεμβαίνει κανείς στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Εμείς στην Δανία, στους νόμους μας, δεν υπάρχει η πρόβλεψη του κατώτατου μισθού. Όμως υπάρχουν κατώτατοι μισθοί σε διάφορους βιομηχανικούς κλάδους. Και όταν γίνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, γίνονται οι υπολογισμοί και η δική μας η μέθοδος υπολογισμού αν τελικά δεχθούμε αυτό που προτείνεται εδώ, ε, θα ήταν αντίθετη με αυτά τα οποία επιβεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Άρα δηλαδή εδώ στη Δανία δεν θα μπορούσε πλέον ε, να υπάρχει μισθολογική πρόβλεψη της τάξης του 50%. Αυτό όμως ε, είναι απαράδεκτο για μας, ε, γιατί δεν είναι δυνατόν να εφαρμόζονται τόσο χαμηλή μισθή. Βεβαίως μπορεί κανείς να πει ή να μιλήσει για ελάχιστο εισόδημα και αυτό μπορεί κανείς να το ρυθμίσει με συλλογικές συμβάσεις ή εθνική νομοθεσία. Εμείς ε, δεν θέλουμε να σας χαλάμε ε, όλο, όλη αυτή την προσπάθεια, αλλά αν περάσει αυτή η διάταξη, ε, τότε θα ε, προκαλούνται πολύ μεγάλα προβλήματα στις βόρειες χώρες. Θα επικρατούσε η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση επεμβαίνει στα μισθολογικά των βορείων κρατών. Βεβαίως και εμείς επιθυμούμε να επικρατεί κάποια τάξη στην μισθοδοσία σε αρκετούς κλάδους. Ήθελα απλά να σας το διευκρινίσω αυτό, να ξέρετε ότι αν υπερψηφίσουμε αυτή τη συμβαστική πρόταση θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες. Και γι' αυτό λοιπόν διρωτώ κιόλας. Τελικά ποιος ε, πρότεινε αυτή τη συμβαστική πρόταση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι για να υπάρξει συμβαστική πρόταση πρέπει να συμφωνούν πάνω από μία ομάδα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον άλλο Τόμας, τον Τόμας Μαν. Εξέχον όσο και ο Τόμας Χάντελ. Εξέχοντες και δύο Γερμανοί πολίτες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χέντελ αναμφίβολα κατέληξε σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και καλή έκθεση και συμφωνώ με πάρα πολλές από τις προτάσεις του. Όμως προφανώς στο θέμα του κατώτατου μισθού ε, δίστανται κατά τι απόψεις μας. Είναι αλήθεια ότι σε 21 από τα 27 κρατημένα υπάρχουν κάποιες τέτοιες ρυθμίσεις. Στη Γερμανία μάλιστα καταβάλλεται η προσπάθεια να προβλέπει το κατώτατο μισθό σε νομικές διατάξεις. Εμείς όμως δεν το θέλουμε αυτό. Δεν θέλουμε να περιοριστούν οι ε, δυνατότητες ε, των κοινωνικών εταίρων. Ε, εξάλλου, ελέγχθη προηγουμένως κάτι τέτοιο ότι πρέπει να υπάρχουν καλέ τομεακέ συμβάσεις. Εμείς στη Γερμανία έχουμε καταλήξει μια πολύ ικανοποιητική λύση. Αν τελικά οι κοινωνικοί εταίροι καταλήγουν σε μια συμφωνία και λένε ε, ισχύει αυτή η συμφωνία, υπογράφουν τη συμφωνία, τη δίνουν στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση την υπογράφει και μετά αυτό είναι, έχει ευρεία α, ισχύ. Και για να υπάρξει αυτή η συμφωνία προϋποτίθεται η εμπειρία, οι ειδικέ συνθήκες, γιατί ξέρετε τι γίνεται, αν τελικά ο κατώτατος μισθός είναι πάρα πολύ ψηλός, αυξάνεται η ανεργία. Ε, δεν μπορεί κανείς να το θέλει αυτό. Μιλήσαμε για διάφορες ερμηνείες. Η Τζιν Λαμπέρτ πολύ σωστά είπε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε ένα σαφή ορισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορούμε και να πλησιάσουν οι διάφορες πλευρές η μία την άλλη. Τροπολογία ας πούμε 38, Τζέικο Κάτσιν ή από τους ε, φιλελεύθερους η 39 ή η δική μου η 40 ε, οδηγούν στην ε, ίσως ε, διαγραφή της ε, πολύ καλής πρωτοβουλίας που οδηγεί στο ότι σε τελική ανάλυση πρέπει να υπάρχουν πρακτικές στα κρατημέλη εφόσον αυτές είναι επιτιμητές. Αυτό βέβαια είναι τελείως διαφορετικό από το να λέμε από εδώ και πέρα ενιαία ρύθμιση. Εγώ με την τροπολογία μου 44 προσπάθησα να καθίσω σαφές ότι πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες οι κοινωνικοί εταίροι. Ε, οι συνθήκες ε, στους διάφορους ε, τομείς πρέπει να είναι ευρέως αποδεκτές. Βεβαίως και ο στόχος για όλους μας είναι ίδιος. Θέλουμε δίκαιη μισθοδοσία, οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν όταν έχουν εργαστεί ε, βεβαίως ε, υπάρχουν τόσες μεγάλες διαφορές ε, στους κλάδους και τους τομείς που πρέπει να επιτύχουμε τη συνένεση των κοινωνικών εταίρων. Άρα δηλαδή εκεί πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας. Και με πολλές άλλες προτάσεις του κύριου Χέντελ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Απλά αυτό που σας ανέφερα. Ο κύριος εισηγητής. Εκτός και αν κάποιος άλλος επιθυμεί να παρέμβει. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν επιθυμεί κανείς το λόγο. Ο εισηγητής λοιπόν. Μισό λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη, μόλις έφτασα από την Ιταλία, δεν ξέρω μέχρι ποιο σημείο έχετε φτάσει, αλλά επειδή είμαι σκιώδης συγγήτρια για αυτή τη γνωμοδότηση από πλευρά ΕΛΚ, θα ήθελα να πω ένα-δυο πράγματα. Δεν ξέρω αν τα είπε ο Τόμας, αλλά θα τα επαναλάβω το πολύ πολύ. Για την τροπολογία 41 και για το συμβασμό C, η άποψη του ΕΛΚ επί του θέματος είναι να απορρίψουμε και τις δύο εκδοχές, και την τροπολογία 41 και το συμβασμό C. Και για το ΕΛΚ είναι πολύ σημαντική ψήφος, γιατί ε, εάν ε, ε, περάσουν αυτά μπορεί να απορρίψουμε και το σύνολο της, της γνωμοδότησης. Ο λόγος είναι απλός. Δεν συμφωνούμε με την εισαγωγή μια συμφωνίας πλαίσιο, μια συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, διότι δεν συμβιβάζεται κάτι τέτοιο με την αρχή της επικουρικότητας και ζητώ συγγνώμη, θα χρησιμοποιήσω ένα επίθετο που ίσως είναι λίγο παραπάνω στεναρό από ό,τι πρέπει, αλλά θεωρώ παράλογο να εισαγάγουμε στοιχεία τη γνωμοδότηση εδώ για θέματα τα οποία συζητήσαμε πριν από δύο εβδομάδες στην έκθεση Φιγκερέιδο και η θέση μας επί των θεμάτων αυτών δεν αλλάζει μετά από δύο εβδομάδες. Αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι πολλές φορές μας προσάπτουν ότι είμαστε πάρα πολύ αργοί στις ε, διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ζητήσω από τους συναδέλφους να μην ακολουθήσουμε αυτή την άγουσα, διότι χάνουμε χρόνο, συζητάμε συνεχώς τα ίδια πράγματα και σε αυτή την περίπτωση Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε ευρύτατα πριν από δύο εβδομάδες και πριν από δύο εβδομάδες στην έκθεση Φιγκερέιδο και πάλι το θέμα αυτό ήταν βασική ψήφος. Και για τον συμβιβασμό ΣΥ λοιπόν και για την τροπολογία 41 η θέση μας είναι να τους καταψηφίσουμε και ε, θα αποτελέσει και βασική ψήφο για την τελική έκθεση. Ένα ακόμα θέμα το οποίο δεν ξέρω αν συζητήσετε αλλά δεν πειράζει η επανάληψη μη τυρμαθήσεως. Η προφορική τροπολογία... entrare ε, ε, in Europa sia legalmente για την ε, έστω και νόμιμη ένταξη των ε, όσων φροντίζουν κάποιους ανθρώπους. Πρόκειται για εργαζόμενους που θεωρούμε ότι είναι στον τομέα της υγείας ε, και της μέρημνας. Και εδώ μπορούμε να έχουμε και νέες παράνομες ε, εισόδους μεταναστών. Ο εισηγητής δεν έχει κατά νου πολύ καλά τι σημαίνει να έχουμε ε, παράνομους μετανάστες ε, στις ακτές της Ιταλίας, της Μάλτας ή κάποιους άλλους οι οποίοι βρίσκονται στη Μεσόγειο, θα ήθελα να σας ζητήσω να έρθετε για διακοπές στη Λαμπεντούσα, να δείτε πώς έχει κατάσταση και αυτές οι τροπολογίες από εκεί και πέρα δεν θα ξαναπροταθούν. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε εισηγητά, να, έχετε πρόσκληση, μπορείτε να πάτε. Σας δίνω το λόγο πάντως για τη συνέχεια της συζήτησης, παρακαλώ. Κοιτάξτε, ε, πρέπει να σας πω ότι σπάνια μένω άφωνος, εννέος, αλλά αυτά που μόλις τώρα άκουσαν με οδηγούν στο να πω σε μία από τις σπάνιες φορές έχω μείνει ενεός. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Όσον αφορά το σημείο υπαριθμών 8, εδώ πρόκειται προφανώς ε, για λάθος ε, εκ παραδρομής, δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τίποτα άλλο, πάντως θα το ρυθμίσουμε και ε, θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα πριν ε, από την ψηφοφορία. Κατάλληλα συμφωνώ με τις επιφυλάξεις σας. Όσον αφορά τα άλλα θέματα, κυρίως αυτά που σε σχέση με τους κατώτατους μισθούς, επιτρέψτε μου να κάνω δύο-τρεις παρατηρήσεις. Συνάδελφε Μαν, εγώ είχα επισημάνει και συνάδελφε Κρίστενσεν, εγώ είχα επισημάνει ότι το θέμα δεν είναι να καταλήξουμε σε μια εθνική ρύθμιση, τομεακή, πολυκλαδική, περιφερειακή. Δεν θέλουμε να αντικαταστήσουμε απολύτως τίποτα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε έστω σε ένα στόχο, ότι η, ε, η φτώχεια οδηγεί σε κατωτατούς μισθούς και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήδη τοποθετήθηκε από και βρήκε μία διατύπωση. Εμένα που δεν είδε με ενδιαφέρει ε, να διαταράξω τις ε, συλλογικές ε, συμβάσεις ή να τα παραγκονίσω τα συστήματα αυτά στα κράτη-μέλη. Εγώ ήμουνα και είμαι ενεργό μέλος ε, του συνδικαλιστικού κινήματος. Ξέρω λοιπόν ε, από το πετσί μου πόσο σημαντική είναι η αυτονομία των ε, συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αλλά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι να πούμε ότι σε όλους τους κλάδους η δύναμη των κοινωνικών εταίρων έχει τόσο πολύ υπονομευθεί που δεν μπορούν πλέον να διαμορφωθούν μισθοί και στην Ευρώπη το καθήκον της κοινωνίας είναι να ορίζει ένα στόχο, να ορίζει το κατώτατο όριο των μισθών, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην διολυσθένουν στην παινία, στη φτώχεια. Αυτό δεν έχει σχέση με την ιδεολογία, αυτό έχει σχέση με το κοινωνικό κράτος πέρα από πολιτικές πεπιθήσεις. Ας πάμε τώρα ε, στις αποχρώσεις που ισχύουν ε, στα βόρεια κράτη ή σε άλλα κράτη. Θέλω να σας πω ότι εμείς δεν επιθυμούμε την επιδείνωση των ρυθμίσεων ο στόχος μπορεί να είναι πολλαπλός και νομίζω ότι είναι θέμα των ε, κοινωνικών εταίρων να επιδιώξουν έναν κατώτατο μισθό ο οποίος είναι υψηλότερος από το κατώτατο κοινωνικό όριο. Αυτά είχα να πω από αυτού του θέματος. Εμείς εργαστήκαμε ουσιαστικά για τους ε, συμβασμούς. Ε, πράγματι μέχρι τώρα ε, δεν έχουμε επιτύχει μεγάλο αριθμό ατόμων που να συμφωνούν με την ε, γνωμοδότησή μας. Ε, σας παρακαλώ να το ξανασκεφτείτε, να δείτε πως έχουμε ουσιαστική υποχρέωση απέναντι στο κοινωνικό κράτος. Για όλες τις άλλες τροπολογίες θέλω να ευχαριστώ όλους όσοι ασχολήθηκαν. Υπάρχουν πολλοί που στηρίζουν αυτές τις τροπολογίες και πέρα από ιδεολογικούς διαχωρισμούς. Θέλω να πιστεύω ότι αύριο θα εγκριθεί η γνωμοδότηση και θα καταλήξουμε σε κοινή απόφαση. Ευχαριστούμε κύριε Σίγητα. Ψηφίζουμε αύριο την γνωμοδότηση αυτή για την Επιτροπή Δικαιωμάτων της Γυναίκας, η οποία από την πλευρά της θα ψηφίσει τέλη Σεπτεμβρίου. Το κείμενο θα πάει στην Ολομέλεια στη δεύτερη σύνοδο του Οκτωβρίου. Και ερχόμαστε στο τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα. Θα σας παρουσιάσω την θέση του Κοινοβουλίου σχετικά με το σχέδιο προπολογισμού 2011, μια που μου αναθέσατε την ευθύνη αυτή. Εγκαινιάζουμε φέτος μια νέα δημοσιονομική διαδικασία, γιατί είμαστε υπό το καθεστώς της συνθήκης της Λισαβόνας. Όπως το είπα και στην αρχή στις ανακοινώσεις μου, γι' αυτό βρισκόμαστε με το ένα πόδι μέσα με το άλλο έξω. Δηλαδή έχουμε το σχέδιο γνωμοδότησης με 14 τροπολογίες, από την άλλη όμως πρέπει να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας με νούμερα. Ακόμα και αν το έγγραφο πάνω στο οποίο αρχίζαμε να δουλεύουμε δεν είναι εκείνο το οποίο επίσημα πρέπει να κρίνουμε δουλέψαμε στο κείμενο της Κομισιόν, ενώ επειδή περνάμε σε συμφωνία με πρώτη ανάγνωση υπό τη Λισαβόνα, πρέπει να αποφανθούμε πάνω στο κείμενο του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο ίσως χαμήλωσε, ίσως αύξησε κάποιες γραμμές σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει ανάλογα να προσαρμόσουμε και εμείς τη θέση μας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας παρουσιάσω το σχέδιο γνωμοδότησης αυτό. Έχουμε 14 προτάσεις για τροπολογίες. Εγώ προσωπικά έχω υποβάλει 9 τροπολογίες, οι οποίες δεν προσθέτουν τίποτα. Οι οποίες καταχρώνται λίγο πολύ από τη διαδικασία τροπολογιών, προκειμένου να αναπτύξουμε παρετέρω κάποια σημεία τα οποία δεν έχουν αναπτυχθεί αρκετά επειδή υπάρχουν οι γνωστοί κανόνε για τι γνωμοδοτήσει, οι οποίε είναι περιορισμένε. Γι' αυτό δεν υπήρχαν στο αρχικό κείμενο αλλά με τη διαδικασία αυτή τροποποίηση έχουμε την ευκαιρία να προσθέσουμε κάτι στο ένα στο άλλο σημείο. Μετά έχουμε τέσσερι τροπολογίε τη κυρία Φιγκερέδο. Η μία έχει να κάνει με τον διπλασιασμό του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για να ανταποκριθούμε στην κρίση. Η δεύτερη είναι για το πρόγραμμα Progress. Η τρίτη είναι για να παραταθούν οι μελέτες για τους αποσπασμένους εργαζόμενους και η τέταρτη έχει να κάνει με την παράταση του πειραματικού προγράμματος όσον αφορά την επισφαλή εργασία. Η κυρία Ίσεν επίσης έχει μία τροπολογία προτείνοντας ένα πειραματικό πρόγραμμα για τους νέους. Όσον αφορά τα νούμερα τώρα, το κείμενο το οποίο δεν είναι επίσημα κοινοβουλευτικό κείμενο ακόμα, έχουμε 32 τροπολογίες. Εγώ προσωπικά έχω καταθέσει 16. 16 τροπολογίες οι οποίες βάζουν ποσά στις προτάσεις της γνωμοδότησης. Στα νούμερα αυτά θα βρείτε τρία νέα πειραματικά προγράμματα καθώς επίσης και την παράταση των προηγούμενων πειραματικών προγραμμάτων που επικυρώνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι προτάσεις αυτές συνάδουν με τις αποφάσεις που έλαβαν οι συντονιστές προς την ίδια αυτή κατεύθυνση. Μία από τις 16 τροπολογίες τέλος προσθέτει ένα νέο στοιχείο το οποίο επιτρέπει να αυξηθεί ο φάκελος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόληση για να ενισχυθεί η μονάδα που ασχολείται με το Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση. Ο στόχος μας είναι, σύμφωνα και με τον κύριο Πόρτας και την κυρία Μωράν, να εξοπλίσουμε τη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση έτσι ώστε να επεξεργάζονται τα διάφορα θέματα πιο γρήγορα, να επιταχυνθούν δηλαδή οι εργασίες. Γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει τεράστια κριτική για αυτό το θέμα, για τις καθυστερήσεις. Αν μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε αυτό το σημείο θα ήταν χρήσιμο. Έχουμε επίσης και 7 τροπολογίες από την κυρία Μπάστος. 6 της κυρίας Φιγκερέδο και μία της κυρίας Ήρς θέλω να μιλήσω για αυτές. Για τις τροπολογίες της κυρίας Βάστος πρώτα. Η πρώτη, δυστυχώς, αντιφάσκει με την τελευταία τροπολογία μου που σας παρουσίασα. Γιατί επειδή υπάρχει οικονομική κρίση, πρέπει να μειώσουμε και τις δαπάνες στο προσωπικό και στη λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόληση, λέει η τροπολογία της. Ακόμα και για το Progress ή για άλλα μέσα στήριξης της προταξιακής διαδικασίας. Αλλά η κυρία Μπάστος από την άλλη μεριά θέλει αύξηση κάποιων ε, άλλων γραμμών στον προπολογισμό. Και στο ίδιο πνεύμα, όπως και η κυρία Φιγκερέιτο και η κυρία Μπάστος, προτείνει να αυξηθεί η γραμμή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με διαφορετικό ποσοστό. Η ίδια τάση πάντως. Η ίδια τάση αύξησης υπάρχει και για την υπηρεσία και την απασχόληση, που ξεπερνάει τις δικές μου προτάσεις. Και υπάρχει και μία πρόταση χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Progress με νούμερα. Για την κυρία Φιγκερέιδο τώρα. Η κυρία Φιγκερέιδο ζητά έψηση για το κοινωνικό ταμείο, Progress ή για τις δράσεις κατάρτισης και επιμόρφωσης υπέρ των οργανώσεων των εργαζομένων. Η τροπολογία της κυρίας Ήρς τώρα αντιστοιχεί στην τροπολογία που περιέγραψα εγώ στο προσχέδιο προπολογισμού και έχει να κάνει με ένα πειραματικό πρόγραμμα για τους νέους οι οποίοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο. Πρέπει να προσαρμόσουμε τις τροπολογίες αυτές στα νούμερα, ανεξάρτητα δηλαδή με ότι ό,τι νέες έχουμε, Χρειάζεται αυτή η προσαρμογή έτσι κι αλλιώς. Η προθεσμία εξάλλου για την των τροπολογιών έχει λήξει, αλλά πρέπει να γίνει προσαρμογή βάσει του κειμένου που θα κληθούμε να ψηφίσουμε, που θα μας έρθει από το Συμβούλιο δηλαδή. Εδώ η Γραμματεία θα μας βοηθήσει βέβαια. Στη συνέχεια υπάρχει ένα έγγραφο που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας επίσης που είναι τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πειραματικά προγράμματα και για τις προπαρασκευαστικές δράσεις που μας ενδιαφέρουν. Θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι εδώ? Ναι. Σε λίγο θα σας δώσω το λόγο. Θέλουν να καταργήσουν κάποια προγράμματα παρά τα σχόλια που πήγανε από εμά και στην Επιτροπή Προπολογισμών και στην ε, Εκτελεστική Επιτροπή και μετά υπάρχουν και κάποιες προτάσεις από ορισμένους ευρωβουλευτές. Καμιά δεκαπενταριά είναι νομίζω. παρουσιάζονται κατευθείαν στην Επιτροπή Προπολογισμών. Έχουμε και ένα πρόβλημα χρονοδιαγράμματος, αλλά αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, θα το δούμε μετά. Καλύτερα να δώσω τώρα το λόγο στην Εκτελεστική Επιτροπή. Να μας πει τη γνώμη της για τα πειραματικά προγράμματα που έχουμε μπροστά μας και μετά θα δώσω το λόγο στους αδέρφους του κ. Μπαστός για παράδειγμα που τη ζήτησε, που ζήτησε το λόγο και σε άλλους. Λοιπόν, Εκτελεστική Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Για τα πειραματικά προγράμματα, η Επιτροπή απάντησε σχετικά με τον μακρύ κατάλογο πειραματικών ε, προγραμμάτων. 19 τέτοια προγράμματα για τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης από τα 150 συνολικά. Χωρίς να πούμε σε λεπτομέρειες, η απάντηση ταξινομεί τη, τα διάφορα αυτά πειραματικά προγράμματα ανάλογα με το πόσο, ε, με τη σκοπιμότητα που έχουν αυτά. Οι απαντήσεις μας αναφέρουν επίσης και την νομική βάση που μπορεί να καλύψει αυτές τις δράσεις. Εκείνο για το όλους Κούβερς. Απαντήσαμε ότι οι δράσεις χρηματοδοτούνται πλήρως από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και ενδεχομένω και από προγράμματα της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΑΚ. Για τα ήδη υπάρχοντα πειραματικά προγράμματα που υπάρχουν πέντε. Για τέσσερα από αυτά κρίνουμε ότι δεν θα ήταν καλό να δώσουμε παράταση αμέσως. Η απάντηση αυτή έρχεται από τις επιχειρησιακές μονάδες, ενώ υπάρχουν προγράμματα που μόλις ξεκινάνε. Γίνεται δηλαδή ο διαγωνισμός. Στα τέλη της χρονιάς θα εγκριθούν, οπότε οι δράσεις λαμβάνουν χώρα το 2011 μόνο. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι ενδιαφέρον να δούμε ποια θα είναι τα πρώτα αποτελέσματα πριν αποφασίσουμε για παράταση και για πόσο. Γι' αυτό και δώσαμε την απάντηση που δώσαμε. Όπως επίσης επειδή η Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης δεν είναι σε θέση να χειριστεί 19 πειραματικά προγράμματα όπως προτάθηκε. Προσπαθούμε να βάλουμε κάποιες προτεραιότητες. Επιτρέψτε μου, παρακαλώ να κάνω και κάποια σχόλια για το τι θα έρθει από το Συμβούλιο, τι να περιμένετε από το Συμβούλιο. Έβαλε μια πρώτη δράση που έκοψε όλες τις πληρωμές, έτσι απότομα. Και την κοινική Διεύθυνση Απασχόλησης περιόρισε τις πιστώσεις για το εντύνιο πάρα πολύ και για τις αυτόνομες γραμμές και για το Progress. Το επίπεδο στο οποίο φτάνουμε τώρα για το Progress είναι τέτοιο που πιστεύουμε ότι είναι δύσκολο να πληρωθούν οι δράσεις το 2011. Για το σόλα κλπ. Οι περικοπές είναι σημαντικές. Πάνω από ένα δισεκατομμύριο. Αλλά πάνω από 200 εκατομμύρια για το ΕΦΣΕ. E. Οπότε βασιζόμαστε στο Ταμείο Συνοχής, στο ΦΕΔ. Η αρχική πρόβλεψη ήταν μια μικρή αύξηση σε σχέση με το 2010. Κάτι άλλο που απασχολεί την Κομισιόν σε σχέση με το τι κάνει το Συμβούλιο είναι για μια διοικητική γραμμή για το προταξιακό μέσο. Το Συμβούλιο προτείνει να κοπούν 10 δισεκατομμύρια στις υποχρεώσεις από τα επιχειρησιακά προγράμματα σε αντίθεση με την πολιετή απόφαση που υιοθετήθηκε τον Οκτώβριο του 2009. Η περικοπή αυτή βάζει τις υποψήφιες χώρες σε μια κατάσταση αβεβαιότητας για το τι λεφτά θα πάρουν ώστε να κάνουν τον πολιτή τους προγραμματισμό και να ετοιμάσουν τις δομές που χρειάζεται για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του κοινωνικού ταμείου όταν θα έχουν ενταχθεί. Από την άλλη το Συμβούλιο έκοψε και την ε, διοικητική γραμμή του προγράμματος ΥΠΑΝ. Η γραμμή αυτή χρησιμεύει κύρια για να δίνει στις αντιπροσωπείες, στις υποψήφιες χώρες, τα μέσα που χρειάζονται για να ελέγχουν, να αξιολογούν και να ελέγχουν οικονομικά τις δράσεις που αναλαμβάνουν υποψήφιες χώρες. Είναι λοιπόν η χρηματοδότηση των τοπικών υπηρεσιών. Πέρυσι με 1,3 εκατομμύρια ευρώ ε, ξοδεύτηκαν τα χρήματα, ενώ τώρα έχουμε 975 εκατομμύρια, κάτι το οποίο μας επιτρέπει να πληρώσουμε ίσα ίσα τους υπαλλήλους εκεί. Και δεν μπορούμε να προβούμε σε υπεργολαβία ή να ζητήσουμε κάποια πρωτογνωμοσύνη για τοπικά προγράμματα. Η πρώτη ανάγνωση περιορίζει τον προπολισμό στα 900.000 ούτε καν το προσωπικό που ήδη υπάρχει. Ε, υπάρχει εκεί το προσωπικό, ούτε αυτό δεν μπορούμε να το πληρώσουμε για τους επόμενους 12 μήνες. Αυτά είναι τα κύρια σημεία που είχα να σας αναφέρω. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, για το progress λέτε ότι το Συμβούλιο μείωσε την προβλεπόμενη γραμμή. Μπορεί, βάσει της συμφωνίας που έχουμε και που εξασφάλισε τη χρηματοδότηση τις πρωτοβουλίες για τις μικροπιστώσεις ή τίθεται υπό αμφισβήτηση. Μόνο για τις πιστώσεις υποχρεώσεων κάνανε περικοπές, δεν μειώσανε... Όχι, μόνο για τις πληρωμές κάνανε, μείωση, όχι για τις υποχρεώσεις. Η κυρία Μπάστος και η κυρία Φιγκερέρο μετά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο που είναι και η συγγήτρια για αυτά τα ε, κονδύλια που προβλέπονται για την απασχόληση για την επόμενη χρονιά. Έχουν κατευθεί τροπολογίες ε, για τις μεμονωμένες γραμμές του προϋπολογισμού που αφορούν στην απασχόληση Εμείς ε, επιθυμούμε ένα άνοιγμα ε, να μπορούμε δηλαδή να υλοποιήσουμε τρία πιλωτικά προγράμματα. Και θα ήθελα να προσθέσω το εξής. Αυτό το έχω πει και κατά το παρελθόν. Εγώ κατέθεσα τροπολογίες με αυτή την έννοια, δηλαδή στη Γενική Διεύθυνση Εργασίας προβλέπεται να καταργηθούν θέσεις απασχόλησης. Και ε, κατ' ουσίαν ε, είχαμε προσθέσει, είχαμε προβλέψει σε γραμμές του προπολογισμού να προσθεθούν κονδύλια, ε, να έχουμε περισσότερες θέσεις εργασίας και διατήρηση θέσεων. Θα ήθελα να πω λοιπόν πιο συγκεκριμένα το εξής. Οι τροπολογίες που κατέθεσα για το 040 41 και 201. Εκεί δεν πρόκειται για την περικοπή των κονδυλίων για ανθρώπινο δυναμικό. Πρόκειται απλά και μόνο για τις διοικητικές δαπάνες που θίγονται. Δηλαδή το θέμα δεν είναι ότι θα υπάρξει κάποια περικοπή. Αυτό που ενδιαφέρει είναι να διατηρηθούν οι θέσεις απασχόλησης και να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε λίγο πιο περιοριστικά στις ε, διοικητικές δαπάνες. Κατά τα άλλα, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προτιμήσουμε εκείνες τις γραμμές του προπολογισμού που ασχολούνται με την απασχόληση. Κυρίως ε, ε, τις γραμμές προπολογισμού που προβλέπουν την πρόθεση της απασχόλησης έχουν σχέση με το κοινωνικό ταμείο. Εκεί επιθυμούμε αύξηση. Το ίδιο ισχύει και για τα πιλωτικά προγράμματα. Προτείνουμε λοιπόν να ε, διατεθούν 2 ε, ε, εκατομμύρια περισσότερα και να ενισχυθεί η κινητικότητα. Εξάλλου, εμείς επιθυμούμε να υπάρξουν την επόμενη χρονιά πιλωτικά προγράμματα με στόχο την προαγωγή της απασχόλησης, κυρίως ε, σε αυτή την περίοδο της κρίσης. Θα ήθελα να αναφερθώ και σε ένα άλλο παράγοντα που έχει σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής ε, στην Παγκοσμιοποίηση. Εκεί ε, προβλέπεται η πρικοδότηση των 50 εκατομμυρίων. όπως αναφέρει και η κυρία Περές στην τροπολογία υποαριθμών 5, αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα για να επιτύχουμε ομαλοποίηση του Ταμείου αυτού. Ε, εμείς ε, στηρίζουμε και την ε, τροπολογία της κυρίας Φιγκερέντο, όπου γίνεται λόγος για τις αλλαγές που πρέπει να λάβουν χώρα στον προπολογισμό. Βεβαίως εκεί γίνεται λόγος για χρήματα. Θα πρέπει να είμαστε λιγάκι πιο μετριοπαθείς για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτά που είναι εφικτά. Καλή είναι η φιλοσοφία, το γνωρίζουμε αυτό, αλλά να ξέρουμε κιόλας ότι δεν υπάρχουν χρήματα και οι προτάσεις ε, να προσθεθούν κονδύλια, ε, όπως προτείνει η κυρία Φιγκερέντο, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο να υλοποιηθεί. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Φιγκερέιδο θα έχει και αυτή την ευκαιρία να στηρίξει τις τροπολογίες της και μετά η κυρία Χίτς. Παρακαλώ κύριε Φιγκερέιδο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και να ευχαριστήσω και τις αγαπητές συναδέλφους που ήδη εξέφρασαν την άποψή τους για τις προτάσεις μου. Ήθελα να πω τα εξή. Όταν αναγνωρίζουμε τα σοβαρά προβλήματα που έχουν οι λαοί των χωρών μας, είτε πρόκειται για ανεργία, είτε πρόκειται για έμβια, είναι λογικό αν θέλουμε να υπάρχει μια κάποια συνοχή μεταξύ των πράξεών μας και των ε, λεγόμενών μας, θα πρέπει να παρουσιάζουμε προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να προσδίζουν κάποια πρακτική ουσία στην επίλυση των προβλημάτων. Έκανα μία απόπειρα εδώ. Να τονίσω, όπως ε, ήδη είπε και η πρόεδρος όταν αναφέρθηκε στις προτάσεις μου, κάποια από τα μεγάλα προβλήματα τα οποία ε, συζητούμε καθημερινά και μάλιστα και σε όλες τις συνεδριάσεις. Σαφώς χρειάζονται χρήματα για να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Αλλά είναι εξίσου σημαντικό οι υπεύθυνοι του προπολογισμού να έχουν μια σαφή εικόνα των προβλημάτων δίνοντας κάποια από τα κονδύλια τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή ακριβώς για να ενισχυθούν αυτοί οι συγκεκριμένοι κοινωνικοί τομεί, συλλαμβάνοντας υπόψη και τη σοβαρή κοινωνική κρίση που βιώνουμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τους τομεί αυτούς ή και να ενισχύσουμε και όλο το γενικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι τούδε δεν έχει τεθεί το θέμα επιτάπητο, αλλά θα έπρεπε να είχε συζητηθεί αυτό το ενδεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη πόσο σημαντική είναι αυτή η κοινωνική κρίση. Οι προτάσει μου δεν είναι ε, θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο, εγώ μπορώ να σας δώσω πάρα πολλά παραδείγματα στα οποία θα μπορούσαμε να ε, βρούμε αυτά τα κονδύλια. Παραδείγματο χάρη, αμυντικές δαπάνες, αν το περιορίσουμε αυτές, σίγουρα θα βρούμε επιπλέον χρήματα. Επίσης, ως προς τα κατόφλια, θα πρέπει να ενισχυθούν κυρίως τα θέματα της απασχόλησης και η καταπολέμηση των διακρίσεων και να γίνουν κάποια πράγματα υπέρ των ίσων δικαιωμάτων και ευκαιριών ε, ε, μεταξύ ανδρών και γυναικών. Αυτοί οι τρεις τομείς είναι πάρα πολύ ευάλωτοι και μέχρι τη δημιουργία του προγράμματος Progress υπήρχαν συγκεκριμένα προγράμματα ε, για κάθε ένα από αυτούς τους τομείς. Κατ' εμέ, ήταν πιο αποτελεσματικά αυτά τα προγράμματα και γιατί συζητήθηκε από πάρα πολλούς ανθρώπους, ενώ με το Progress δεν ισχύει το ίδιο. Εδώ βέβαια το πρόβλημα είναι τα χρήματα. Αυτό που έκανε το Συμβούλιο είναι απαράδεκτο. και όχι μόνο για τους κοινωνικούς αυτούς τομείς ε, στους οποίους αντιμετωπίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Ε, έγιναν ε, περικοπές ε, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως ε, την περσινή χρονιά, αλλά όλα αυτά δεν μας επιτρέπει να, επιτρέπουν να προοδεύσουμε και να δώσουμε μια απάντηση στο μέλλον. Οι προτάσεις μου λοιπόν για το progress είναι καθόλου δικαιολογημένε σε αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον και όλα όσα έχουν να κάνουν με το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο δικαιολογούνται. Αυτά θα πρέπει να τα δούμε όχι μόνο υπό το πρίσμα του κατά πόσο χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και μια νέα οπτική γωνία που έχει σχέση με την έκθεση που συζητούμε αυτή τη στιγμή για το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα ε, για την καταπολέμηση της φτώχειας. Θεωρώ ότι είναι υψής της σημασίας να υπάρχει ένα μέσο στον προϋπολογισμό το οποίο θα μπορέσει να απαντήσει στο πρόβλημα της ένδυας. Και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα από τα μέσα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ακριβώς προς αυτό το σκοπό. Ο Επίτροπος ε, αναγνώρισε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα μπορούσε να διαδραματίσει πολύ σημαντικότερο ρόλο στην αντιμετώπιση της φτώχειας και εγώ σε αυτό αναφέρομαι. Κάνω μία πρόταση η οποία σαφώς δεν επιλύει το πρόβλημα της μιζέριας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα μπορούσε να είναι ένα χρήσιμο μέσο για να μπορέσουμε να την ε, μειώσουμε την ένδυα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σαφώς ισχύει. Υπάρχουν δράσεις κατάρτισης, ε, υπάρχουν δράσεις κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της ένδυας και όλες αυτές οι δράσεις θα μπορούσαν να είναι ολοκληρωμένες και να κατευθύνονται, να απευθύνονται στους φτωχούς που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Δεν νομίζω ότι χρειάζονται περαιτέρω εξηγήσει. Νομίζω ότι οι προτάσεις μου επικεντρώνονται ακριβώς ε, στην επίτευξη αυτών των μεγάλων προκλήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Merci, Madame Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω ε, που είστε εισηγήτρια και για την τροπολογία υπαριθμών 9, όπου στοχευμένα αναφέρεται ότι οι ευκαιρίες για τους ε, νέους ε, να βρουν απασχόληση, αυτό είναι προτεραιότητα και ως εκ τούτου αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και σε ένα προϋπολογισμό. Νομίζω είπατε με απόλυτη σαφήνεια ότι είναι προτεραιότητα, αυτό το βλέπουμε επανειλημμένα, έχουμε συστήσει επανειλημμένα το θέμα της ανεργίας ε, στην Επιτροπή μας και διαπιστώνουμε ότι η ανεργία των νέων αυξάνεται. Τρομάζει το να βλέπει κανείς ότι πολλοί άνθρωποι, πολλοί νέοι ε, που έχουν σπουδάσει, που έχουν ε, τελειώσει το σχολείο παραμένουν άνεργοι Γι' αυτό λοιπόν αυτή η ε, τροπολογία αφορά ε, κυρίως τους ανθρώπους που διακόπτουν τις ε, σπουδές τους οι άνθρωποι αυτοί να κινητοποιηθούν, να βρουν απασχόληση, γιατί εγώ ανησυχώ. όταν βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν, όπως σας είπα, κάποια προσόντα, σχολείο, σπουδές, αυτοί το να είναι άνεργοι Καταλαβαίνετε πόσο μάλλον οι άνθρωποι που έχουν διακόψει το σχολείο ή τις σπουδές τους, αυτοί είναι σε τραγική μοίρα. Αυτοί, για αυτούς είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρούνε εργασία. Στην ε, Στρατηγική Ευρώπη 2020 είπαμε με σαφήνεια ότι θέλουμε να περιορίσουμε τον αριθμό των νέων που διακόπτουν ε, το σχολείο. Ε, Παρ' όλα αυτά θα υπάρχει ένα σημαντικό ποσοστό που θα έχει εγκαταλείψει το σχολείο. Άρα δηλαδή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει ένα ευδιάκριτο μήνυμα ε, να αναφερθούμε σε αυτούς τους ε, ανθρώπους, να ξεκινήσουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα και να πούμε ότι νέοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δυνατότητες. Ίσως να μην τα κατάφεραν στο σχολείο, όμως έχουν δυνατότητες και με αυτούς τους ε, νέους μπορούμε να δουλέψουμε, να τους προσφέρουμε μια ευκαιρία, ίσως σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις. Βεβαίω, ε, τέτοιο ερώτημα κατά πόσον αυτά τα προγράμματα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το κοινωνικό ταμείο. Αν δείτε όμως τα προγράμματα αυτά, βλέπετε ότι αφορούν νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια εκπαίδευση. Άρα δηλαδή, ε, στόχευμένα πρέπει να προβάλλουμε αυτήν την ομάδα των νέων να πούμε ότι θέλουμε να τους εντάξουμε σε ένα δίκτυο επιχειρήσεων. Αυτό είναι ο στόχος, να συστήσουμε δίκτυο επιχειρήσεων ε, όπου οι νέοι θα γνωρίζουν ότι μπορούν να ενταχθούν εκεί. Να τους πούμε λοιπόν ότι ξέρετε, εμείς ξέρουμε και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να χαθούν. Ελπίζω η Επιτροπή ε, να δώσει ένα ευκρινές μήνυμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Θα έρθω σε επαφή μαζί σας για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Βλέπω βέβαια και κάποιες αντιφάσεις που πρέπει να λυθούν. Για το θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόληση, για την κινητοποίηση των πόρων, για την ε, προσαρμογή στην παγκοσμιοποίηση, με την κυρία Μπάστος πρέπει να βρούμε μια συμφωνία. Γιατί βλέπετε ό,τι και να κάνουμε, είμαστε σε περίοδο δημοσιονομικής λιτότητας. Κανένας δεν θα ξεπεράσει πλήρως την κατάσταση αυτή. Όμως πρέπει να βοηθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν ψηφίσαμε την έκθεση της κυρίας Μωράν, Όλοι είπαν ότι θέλουν την παρέμβαση του Ταμείου αυτού. Από ευρωπαϊκή άποψη, αλλά και από άποψη κρατών μελών, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να έχουμε ένα ευρωπαϊκό μέσο, χωρίς όμως να μπορούμε να προχωρήσουμε με τις φιλοδοξίες μας. Και σήμερα στη Γενική Διεύθυνση Απασχόληση αυτό συμβαίνει. Δεν υπάρχει δυνατότητα παρέμβασης ώστε οι αιτήσει που υποβάλλονται να επεξεργάζονται σε ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα και να υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα. Για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων θα δούμε τώρα τι θα γίνει στο Συμβούλιο. Εμείς όμως ξέρουμε τι διακυδεύεται εδώ. Δεν μπορούμε και εδώ να έχουμε από τη μια την ομάδα εργασία, τη οποία προεδρεύει ο Φαν Ρομπά, ο οποίο ανησυχεί για τι διαφορέ στην ανταγωνιστικότητα των κρατών μελών, να θεωρούμε ότι τα θέματα τη απασχόληση πρέπει να θεωρούνται σαν μια ανισορροπία που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά να μειώνουμε τα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Εμείς ξέρουμε ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ σοβαρό. Υποπολαπλασιάζεται το αποτέλεσμα δηλαδή. Οπότε θα στραφώ προς εσάς για να βρούμε ένα καλό κατάλογο για την ψηφοφορία. Με έναν όσο γίνεται μεγαλύτερο κοινό παρονομαστή. Ευχαριστώ όλους ιδιαίτερως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το έγγραφό της. Είναι πρώτη φορά που έχουμε τόσο συγκεκριμένες απαντήσεις και τόσο ξεκάθαρες. Έτσι ξέρουμε ποια θα είναι η προσέγγιση της Επιτροπής στα θέματα πιλωτικών προγραμμάτων. Αυτό το πνεύμα συνεργασίας που επιδεικνύεται είναι πολύ σημαντικό για μας. Τέλος, οι διορθώσεις, οι τεχνικές τροπολογίες, πώς να το πω, για να έχουμε υπόψη μας τα νούμερα του Συμβουλίου. Μπορεί να μην χρειαστούν αλλαγές, αλλά μπορεί και να πρέπει. Εκτός από αυτό μένει ένα μικρό ερωτηματικό που είναι το χρονοδιάγραμμα. Η Επιτροπή Προπολογισμών δεν είναι ικανοποιημένη από το δικό μας το χρονοδιάγραμμα. Θεωρεί ότι εφόσον εγκρίνουμε το κείμενο στις 13 Σεπτεμβρίου, είμαστε εκτός προθεσμίας, έτσι όπως την καθόρισε η Επιτροπή Προπολογισμών για τις τροπολογίες. Εμείς ζητάμε παράταση και τι έγινε, μας την αρνήθηκαν. Θα δούμε. Μήπως παρόλα αυτά μπορούμε και εκτό προθεσμία να υποβάλουμε τι τροπολογίε μα. Ή μήπως πρέπει να συνεδριάσουμε εκτάκτος τον Σεπτέμβριο στο Στρασβούργο, στην πρώτη σύνοδο. Μου λένε ότι δεν γίνεται, είμαστε οι τελευταίοι που ζητάμε κάτι. Τέλο πάντων, θα δούμε. Πρέπει να βρεθεί μια λύση, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ μέσω ταχυδρομείου εγώ να γκρίνω τον προπολογισμό ή που θα έχουμε μια σύντομη συνεδρίαση, μια έκτακτη σύντομη στο Στρασβούργο η Επιτροπή Προπολογισμού θα πρέπει να δεχτεί τις τροπολογίες μας και σε έχει λήξει η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών. Έτσι καλλιώς 28 με 30 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουν αυτοί. Σα ευχαριστώ για όλα. Τελειώσαμε λοιπόν με τη σημερινή μα ημερήσια διάταξη. Ραντεβού αύριο το πρωί στι 9 για ανταλλαγή απόψεων με τη Βελγική Προεδρία που εκπροσωπείται από την Ζωέλ Μιλκέ που είναι αντιπρόεδρος απερχόμενη για την ισότητα και τις κοινωνικές ε, υποθέσεις και την κυρία Λορέτ Όγενλεξ και τον κύριο Νταρντέν. Ευχαριστώ.